Good morning, everyone. Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ που λάβατε θέσεις και ετοιμάσατε φαντάζομαι τις ηλεκτρονικές κάρτες ψηφοφορίες για να ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες μας αμέσως. για να ολοκληρώσουμε ώστε στις 11 να ξεκινήσουμε την ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο. Επαναλαμβάνω, έχετε όλοι μαζί σας τις ηλεκτρονικές κάρτες ψηφοφορίας. Θα κάνουμε έναν ηλεκτρονικό έλεγχο πρώτα. Uh, σημείο πρώτο, έγκριση της ημερήσεις διάταξης. Συμφωνείτε? Δεν βλέπω σχόλια, οπότε εγκρίνεται. Ανακοινώσεις. Έχω καμιά δυο. Θα έχουμε έκτακτη συνεδρίαση στο Στρασβούργο τη Δευτέρα 13 Μαρτίου, 7 το απόγευμα με 8.30. Θα έχουμε ανταλλαγή απόψε με τον Επίτροπο Αρίας Κανιέτε στα πλαίσια του διαρθρωμένου διαλόγου. Δεύτερη ανακοίνωση, μία αλλαγή στη γραμματεία μας. Η κυρία Ιωάννα Πόστου, διοικητική υπάλληλο, προσχωρεί στη γραμματεία της Επιτροπής Περιβάλλοντος από την 1η Μαρτίου και θα ήθελα να την καλωσορίσω στην Επιτροπή μας. Διερμηνία έχουμε σε 21 γλώσσες με εξαίρεση τρεις. Εστονικά, λιθονικά και βοεδελικά. και έχετε και ηλεκτρονικά τα θέματα μέσω της ε, εφαρμογής e-meeting. Έχετε λάβει και τις ε, συστάσεις των συντονιστών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ελπίζω να τις μελετήσετε και αν δεν ε, υποβληθούν παρατηρήσεις θα θεωρηθούν ως συγκεκριμένες. Επίσης, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, να εγκρίνουμε και τα πρακτικά των συνεδριάσεων της 8ης Δεκεμβρίου και 23, 23ης και 24ης Ιανουαρίου. Θα θεωρηθούν ως συγκεκριμένα αν δεν υποβληθούν προτάσεις ή παρατηρήσεις στη γραμματεία. Περνάμε στις ψηφοφορίες τώρα. Η πρώτη έκθεση είναι η έκθεση Τανασέσκου. Ξεκινάμε με την τροπολογία 57. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αλλά ας κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο γιατί βλέπω διάσπαση σε ορισμένες ομάδες. Τροπολογία 57. Ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 58. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 59. Τροπολογία. Θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο και για την 58. Ο, εντάξει. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 58. Τέλος ψηφοφορίας. ισοπαλία αλλά απορρίπτεται. Τροπολογία 59. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 60. Τροπολογία σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται τροπολογία 9 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 61 υπέρ ε, καταπίπτει συγγνώμη τροπολογία 62 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 11 υπέρ καταπίπτει. Η 11 καταπίπτει. Όχι. Ψηφίζουμε και την 11. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 66 υπέρ κατά αποχές να σηκώνετε τα χέρια σας για να βλέπουμε. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Α, γι' αυτό δεν σηκώσετε τα χέρια. Τώρα μας πρέπει να ψηφίσετε. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνατε. Τροπολογία 70. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 79 υπέρ Θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο για την 78. Ωραία. Άρχεται η ψηφοφορία. Αλλά δεν σηκώνετε τα χέρια σας. Γι' αυτό είναι δύσκολο να δούμε με ανάταση της χειρός αν πέρασε μια τροπολογία. Ε, απορρίπτεται 79 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 80 υπέρ, κατά, αποχές, Ηλεκτρονικός έλεγχος και για αυτήν. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 16. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 81 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 82 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 86 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 89 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος The vote is open The vote is closed Τέλος ψηφοφορίας Adopted ε, Εγκρίνεται 90 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται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 κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 99 υπέρ κατά αποχές Δεν είδα πώς ψήφισαν οι σοσιαλιστές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 99. Άρχεται η ψηφοφορία και τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 100. Υπέρ. Υπέρ της τροπολογίας 100. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 101. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 102 καταπίπτει 104 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 105 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 107 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τις 108 και 109 μαζί υπέρ, κατά, αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τις τροπολογίες 108 και 109 άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. Τροπολογία 110 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 111 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 112 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 113 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 114 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 27 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 115 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 117 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 118 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 28. Καταπίπτει. Εκατόν δεκαεννέα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 120 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 121 υπέρ. Κατά αποχές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 εγκρίνω, εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και 56 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται τελική ψηφοφορία ονομαστική άρχεται ψηφοφορία και τέλος της ψηφοφορίας εγκρίνεται Next vote. Η επόμενη ψηφοφορία αφορά την έκθεση Γκαμπούς. Ξεκινούμε με την πρώτη τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παριθμόν 2. Συμβαστική υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 97. 98 γιατί καταπίπτει 97. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 101 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 103 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτωται. 104 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτωται. 105 υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος για το 105. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Πέρα ψηφοφορία, ναι, εγκρίνεται με σαφή διαφορά ψήφων υπέρ. 106 υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται. 120 υπέρ κατά αποχέ, απορρίπτεται. 6 υπέρ κατά. Ποιοι είναι κατά για το 6. Αποχές εγκρίνεται 107. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται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 κατά αποχές απορρίπτεται 110 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά υπέρ για το 16 κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 20 υπέρ ηλεκτρονικός έλεγχος για το 19. Ψηφίζουμε. Α, έκανα λάθος. Πεςτε μου αν κάνω λάθος μέσα αυτή η πλειοψηφία εγκρίνεται ένα λάθος λάθος λέξη διάλεξα 20 18 18 έλεγχος για το 18 Ψηφίζουμε. 18. Πέρας. Απορρίπτεται. 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 6. Συμβιβαστική. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 118. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 20 27, 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 10. 30, συγγνώμη. 30 εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 113 υπέρ. Σχόλιο εκτός μικροφώνου. Θέλετε να κάνουμε για το 48 ηλεκτρονικό έλεγχο. Μα πού είναι το 48. Ποιο το 28. Πάει αυτό. Το έχουμε πει εδώ και πολλή ώρα. Κάποιες πολιτικές ομάδες δεν, δεν τηρούν ενιαία γραμμή. Αλλού ψηφίζουν το ένα, αλλού το άλλο. Γι' αυτό μπορεί να φαίνεται ότι δεν σας τα λέω κι εγώ με συνέπεια, αλλά... Τέλος πάντων, 113. Υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32. Υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για το 32 ψηφίζουμε και πέρα στις ψηφορίες Α, απορρίπτεται 33 υπέρ κατά αποχές έλεγχος Η Άλντε μου κάνει τη ζωή δύσκολη, λέει πρόεδρο. Πέρα εφορία. Και εγκρίνεται. 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχο Ψηφίζουμε και πέρας ψηφορίας απορρίπτωται Συμβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 36 υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 38 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται συμβαστική 9 εγκρίνεται 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 117 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 42 υπέρ κατά αποχές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 Απορρίπτωται. 54 υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτωται. 55 υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτωται. Συμβαστική 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτωται. 4 in favor, against, abstentions. 64 υπέρ, κατά, απορρίπτωται. 65 υπέρ, κατά, Αποχέ. εγκρίνεται 66 υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 70 υπέρ έλεγχος για το 69 Πέρας. Εγκρίνεται. Αργήσατε να σηκώσετε τα χέρια σας. Μόνο έτσι εξηγείται. Αλλιώς η διαφορά ήταν σαφής. Amendment 70. Το 70 ποιοι είναι υπέρ. Against. Abstention. Κατά αποχές απορρίπτεται. 71 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 76 υπέρ αποχές εγκρίνεται 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτω 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτω 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτωται 82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτωται 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτωται 84 υπέρ κατά αποχές απορρίπτωται 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 86 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 91 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται The vote is open and please vote Ψηφίστε παρακαλώ Πέρας ψηφοφορίας. Και εγκρίνεται και συγχαρητήριο. Επόμενο. Next vote is uh, report. Palm oil. Έκθεση Κονέτσνα για το φινικέλαιο. Ψηφίζουμε καταρχάς DV1 μέρος 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. DV1 μέρος 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ίντα μέρος 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 2 η καταπληκτή. Άγκρι 68 μέρος 1 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Άγκρι 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 6 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 75 ψήφι πέρα κατά αποχές εγκρίνεται. Είναι τα δύο πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Είναι τα πέντε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ντέβε δέκα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική ένα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ. Έχουμε και μια της άγκρη πριν. Α, δεν κατάλαβα, Νόμως ήταν ε, κεφαλίδα. Άγκρη 32 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 87 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 96 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 95 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 97 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 98 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, συμβιβαστική 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 107 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 110 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 113 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 115 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 55 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 132 λέγε υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. ΔΒ11 μέρος 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 140 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 142 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Είναι τα 15, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. ΔΕΒΕ 17 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 159 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 162 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ, κατά, αποχές εκρίνεται Συμβιβαστική 9 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 52 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 186 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 187 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 191 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 201 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 108 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύε 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ίντα 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 128 δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Δεύτερο είναι της 128. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίθηκε. τόσο συγγνώμη. Άκρη 29. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο 23 Δεύτερο τμήμα υπέρ. Όχι. Δεύει 25 πηγαίνουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύε 2. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύε 3. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 67 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 69 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 209 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 12 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 14 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 219 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 15 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 227 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 2.45 υπέρ. Καταπίπτει. Πάμε στο 126 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. ΔΕΒ 24 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. ΔΕΒ 26 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύε 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται μάλλον, αλλά ας ελέγξουμε. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύε 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Όχι, εγκρίνεται. Δεύε 5 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άγκρι 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άγκρι 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύε 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύε 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άγκρι 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 99 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 27 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 8 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 200 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 234 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Άγκρι 70 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δέβε 14 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 18 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 247 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 111 υπέρ, όχι. Έχει καταπέσει, συγγνώμη. Άγκρι 50 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 248 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 34 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 36 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 19 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύε 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Είπα τρίτο τμήμα ότι ήταν. Δεν το είπα, δεν πειράζει. 114 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άκρη 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άκρη 43 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. τα 62 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2,60 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τι είπατε? Κάποιος μιλάει. Ποιος είναι αυτός που μιλάει? Δεν κατάλαβα τι είπατε. Στο μικρόφωνο παρακαλώ να τα λέτε. Θέλετε να ελέγξουμε την άκρη 62. Μάλιστα, οκ, okay, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τώρα πηγαίνουμε στην 260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 απορρίπτεται. 21 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε. Έλεγχος για την 21. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 όχι 33 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε την 33 αρχιτή ψηφοφορία 33 ψηφίζουμε, εντάξει. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνθηκε. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Καλύτερα να ελέγξουμε. 35. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Συμβιβαστική 22 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 23 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συνεργαστική 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, να υποθέσω. Σχεδόν κανένα χέρι δεν σηκώθηκε, δεν πάνω. 55 ελέγχουμε. Πέρασε. εγκρίνεται 51. Καταπίπτει 51. 54 πηγαίνουμε. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 52. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 25, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 59, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 60, υπέρ, Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 69 εντάξει ελέγχουμε την 69 Έληξε ψηφοφορία εγκρίνεται. 70 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 71 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 72 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 73 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 74. Τι κάνουμε, την ψηφίζουμε, την ψηφίζουμε. 74 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ονομοδότηση Επιτροπή ΣΥΝΤΑ τώρα. αυτά δεν τα ψηφίζουμε. Α, ωραίο νέο αυτό. Άρα που πηγαίνουμε στην τελευταία σελίδα και στην τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά παρακαλώ έρχεται ψηφοφορία. Πολύ ευχάριστη έκπληξη αυτή. Περιμένω να ψηφίσετε όλες και όλοι, εφόσον βεβαίως το επιθυμείτε, πέρας ψηφοφορίας. Τουλάχιστον συμφωνήσαμε. Ευχαριστούμε, εγκρίθηκε. Σας ευχαριστώ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ώρα των ψηφοφοριών. Συγχαρητήρα σε όλους. In five minutes uh, we have uh, Commissioner Vela, so don't go far. Μην πάτε μακριά γιατί έχουμε τον Επίτροπο Βέλα.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

So, συνάδελφοι, καθίστε, λέει η Πρόεδρος. Και καλώ ορίστε μαζί μου τον Επίτροπο κύριο Βέλλα. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Ήταν ε, καλοσύνη του που αποδέχθηκε την πρόσκληση ο κύριος Επίτροπος στα πλαίσια του διαρθρωμένου διαλόγου όπως προβλέπετε. Παρακαλώ συνάδελφοι. Ησυχία. Και σας ευχαριστώ. Καλώς ορίζατε, κύριε Επίτροπε. Περιμένουμε πώς και πώς να ακούσουμε μας λέτε για το πρόγραμμα εργασίας του 2017, τις προτεραιότητές σας και είμαι βέβαιος ότι ενδιαφέρονται πάρα πολλοί συνάδελφοι να ακούσουν τι έχει να μας πείτε για τα διάφορα θέματα του θεματολογίου σας για το κοντινό μέλλον. Εδώ θα βάλω τελεία και πάλι καλώς ορίσατε. Έχετε το λόγο. Thank you. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ. Αντίνα, αξιότιμη ευρωβουλευτέ. Τέτοιου είδου ανταλλαγέ απόψεων είναι πραγματικό ορόσημο στο πρόγραμμά μου και έχοντας διατελέσει για ολόκληρες δεκαετίες ε, βουλευτής εθνικός, 38 χρόνια, θεωρώ τέτοιες ανταλλαγές ως ε, σημαντικό τμήμα της λογοδοσίας των δράσεών μας. Ειλικρινή συζητήσει περί πρόοδου είναι εξαιρετικά χρήσιμε και εκτιμώ ιδιαίτερω την ευκαιρία που μου δίνετε να σα κάνω μια ενημέρωση για το τι μπορεί να περιμένετε του επόμενου μήνε. Βρισκόμαστε στο μισό τη ε, θητεία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουν περάσει δύο, δυόμιση χρόνια από τότε που έχω αναλάβει τη θητεία μου, που για πρώτη φορά συνδυάζει το γαλάζιο με το πράσινο, το περιβάλλον, τη θάλασσα και την αλία σε ενιαίο χαρτοφυλάκιο. Μάλιστα αυτός ο συνδυασμός ε, πάει πολύ καλά. Ο συνδυασμός της θάλασσας, της ξηράς και των ωκεανών ε, με την ε, στεριά μας οδήγησε σε μια πιο κοινή προσέγγιση σε συνδυασμό με την κυκλική οικονομία, τα πλαστικά και τα θαλάσσια απορρίμματα, το ρόλο των ωκεανών για το περιβάλλον ή το πώς ε, η βιοπικιλότητα της θάλασσας μπορεί να υποφεληθεί από την καταπολέμηση της παράνομης αλίας. Πριν από λίγες μέρες, ο πρόεδρος Γιούνκερ σας παρουσίασε το πιστοποιητικό γέννηση του μέλλοντος της Ευρώπης, ο προεδρος γιουγκερ σας παρουσιασε το πιστοποιητικο γεννηση του μελλοντος της ευρωπης δηλαδη τη Λευκή Βίβλο που θα ξεκινήσει μία συζήτηση ε, για το μέλλον της Ευρώπης. Ήταν πολύ χρήσιμο το μήνυμα και πολύ ρεαλιστικό. Να κάνουμε ό,τι ε, δουλεύει και μάλιστα ό,τι δουλεύει καλά και αποφέρει καρπούς. Και μάλιστα οι περιβαλλοντικές μας πολιτικές θα πάνε πολύ καλά. Υγούμαστε σε παγκόσμιο επίπεδο, κάτι που μας το ζητάει και συνθήκη, και εξασφαλίζουμε υψηλό επίπεδο προστασίας των πολιτών μας και βελτιώνουμε τη ποιότητα του περιβάλλοντος. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι εξασφαλίζουμε επίπεδα προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι όνειρο άλλων ε, πολιτών, άλλων ε, περιοχών του πλανήτη. Έχουμε καθαρότερο νερό, καθαρότερο αέρα, ασφαλέστερα προϊόντα και αυτό χάρη στη συνεργασία και τη συμφωνία μας. Και 27 χώρες μέλη θα συνεχίσουν να το κάνουν και θα συνεχίσουμε να δίνουμε το καλό παράδειγμα. Από κοινού, μάλιστα, έχουμε ηγηθεί παγκοσμίω στην πρόθεση της ε, κύκλικης οικονομίας. Και θα πρέπει να διαρρήξουμε την ιδέα που υπάρχει και να καταρρύψουμε την ιδέα που υπάρχει ότι η περιβαλλοντική πρόοδος περιορίζει την οικονομική και κοινωνική ευημέρεια. Θα αποδείξουμε το αντίθετο. Και μάλιστα σε λίγες μέρες θα δώσετε εντολή στον εισηγητή σας στην Ολομέλεια να διαπραγματευτεί προτάσεις για να αξιοποιήσουμε οικονομικά τα απόβλητά μας και με ένα χρόνο μετά την υποβολή των προτάσεων είμαι εντυπωσιασμένο από την ταχύτατη πρόοδο που σημειώσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συγχαρητήρια στη Σιμώνα Μποναφέ και στου κοιόδη ηγητέ, γιατί κατέληξαν σε μια ξεκάθαρη στάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι το απόσταγμα περίπου 2.000 τροπολογιών. Η έγκριση των προτάσεων αυτών θα σημάνει ότι αντί να καίμε ή να θάβουμε πολύτιμε πρώτε ύλε στο έδαφο, αναπτύσσουμε αγορέ για τα υλικά αυτά προωθούμε νέα επιχειρηματικά μοντέλα και δημιουργούμε θέσεις απασχόλησης στην κυκλική οικονομία. Και μάλιστα η κυκλική οικονομία περνάει από τα λόγια στα έργα, από τη θεωρία στην πράξη, από τα έγγραφα στην πραγματικότητα, με πολλές πρωτοβουλίες για την πρόωθηση επενδύσεων, για τη χορήγηση των πραγματικών αναυσμάτων και την πραγματοποίηση αλλαγών. Και μάλιστα, όπως μας ε, ε, ζητήσατε, θα δημιουργήσουμε και ένα πλαίσιο παρακολούθησης για να καταμετρούμε την πρόοδό μας στο σχέδιο δράσης της κυκλικής οικονομίας και να παρακολουθούμε την εφαρμογή όλων αυτών των πρωτοβουλειών. Τον Ιανουάριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ενημέρωση της ε, νομοθεσίας για τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές. Και χαίρομαι ιδιαίτερος που η Αντίνα Βαλεάν έχει αναλάβει την ευθύνη και θα εκπονήσει τη σχετική έκθεση. Επίσης εγκρίναμε μία ανακοίνωση για τον ε, ρόλο των αποβλήτων ε, σε σχέση με την ενέργεια στην κυκλική οικονομία, δίνοντας κατευθυντήριες γραμμές στα κράτη-μέλη και τους επενδυτές. Και σημειώνουμε θετική πρόοδο, αλλά δεν προχωρούν όλα τα θέματα της ε, κυκλικής οικονομίας με την ίδια ταχύτητα ή προς την ίδια σωστή κατεύθυνση. Προσοχή λοιπόν, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το θέμα των λοιπασμάτων με σωστό τρόπο. Έχουμε ξεκάθαρα επιστημονικά πορίσματα για τους σημαντικούς κινδύνους και τις ζημίες που μπορούν να προκαλέσουν τα πλαστικά πολυμερή και το κάδμιο στα προϊόντα λίπανσης. Ακόμη και προϊόντα που φέρουν το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υποτίθεται ότι πρέπει να καθησυχάζει τους ανθρώπους έχουν τέτοιο πλαστικά και κάδμιο. Η νέα πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον κανονισμό για τα λιπάσματα ε, σημειώνει, ε, δίνει σημαντικά και απαραίτητα κατόφλια περιορίζοντας το κάδμιο και τα πλαστικά και τη ρήπαση τους ε, τη ρήπαση του εδάφους από αυτά. Και με την αιγίδα της ε, Επιτρόπου Μπιενκόφσκα ήδη προβλέπουμε πολύ λογικές περιόδους ε, σταδιακής εισαγωγής περίοδο ε, το, το, της μείωσης του καδμίου για μία δωδεκαετία, παρόλο που τεχνολογικές λύσεις είναι ήδη διαθέσιμες στην αγορά από σήμερα. Και έχουμε τεράστιες ευκαιρίες για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που θα πρέπει να υιοθετήσουν καλύτερες προσεγγίσεις και να ηγηθούν στην προσπάθεια αυτή στην αγορά. Θέλουμε συνοχή για να υλοποιήσουμε την ε, κοινή μας δέσμευση, να περιορίσουμε τα πλαστικά στο έδαφος, ε, το νερό και το θαλάσσιο περιβάλλον. Και με το νέο κανονισμό για τα λοιπάσματα δεν θα πρέπει να υποβιβάσουμε τις προδιαγραφές ε, του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό σας θέλω παρακαλώ, εξετάστε προσεκτικά τα επιστημονικά πορίσματα που αποτελούν τη βάση της ε, πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ευελπιστώ ότι θα μπορώ να υπολογίσω στη δική σας συνδρομή ώστε να διαφυλάξουμε τα υψηλά μας περιβαλλοντικά πρότυπα και τις υψηλές μας προδιαγραφές όπως περιμένει και ο κόσμος από εμά. Ο ρόλος σας ε, ήταν κέριο σε όλα αυτά τα θέματα της ε, κύκλικης οικονομίας. Λίγο νωρίτερα σήμερα το πρωί κήρυξε τα εγγένεια στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της διάσκεψης των ενδιαφερομένων για την κυκλική οικονομία. Και μάλιστα οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν αύριο στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Η συζήτηση θα εστιαστεί στην μορφή που θα πάρει η πλατφόρμα των ενδιαφερομένων ε, της κυκλικής οικονομίας και θα ήθελα να διαδραματίσετε και εσείς κέριο ρόλο από κοινού με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών. Η κυκλική οικονομία φέρνει κοντά ε, τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, τους ε, επενδυτές και τους επιχειρηματίες, αλλά έχει και μια πολύ σημαντική ανθρώπινη πτυχή. Γιατί η αξιοποίηση των πόρων της ευρωπαϊκής ε, οικονομίας σημαίνει περισσότερες θέσεις απασχόλησης, αλλά θα αλλάξουν και οι θέσεις αυτές, αλλά και οι δεξιότητες που απαιτούνται. Γι' αυτό και στα τέλη Μαΐου θα δημιουργήσουμε την Πράσινη Εβδομάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να παρουσιάσουμε το δυναμικό των πράσινων θέσεων απασχόλησης σε όλους τους τομείς χάρη στην κυκλική οικονομία. Και θέλουμε να μεταβιβάσετε αυτό το μήνυμα και σε εκλογικές σας περιφέρειες για να αποδείξουμε στον κόσμο ότι υπάρχει ένα μέλλον σε όσους έχουν δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην κυκλική οικονομία. Επίσης, θα πρέπει να αποδείξουμε ότι η μέλημά μας είναι να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών με την νομοθεσία μας. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ένα υψηλό βιωτικό επίπεδο και μια ποιότητα ζωής. Αυτό θα πρέπει να το ξεχνούμε κατά την πρόταση, διαπραγμάτευση και εφαρμογή της νομοθεσίας μας. Και μια περίτρενη απόδειξη και χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτών είναι η ποιότητα του αέρα. Η κακή ποιότητα του αέρα είναι ένας αθόρυβος και αόρατος δολοφόνος, αλλά χάρη στις δράσεις μας ε, καταφέραμε οι κυβερνήσεις να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη αυτό το θέμα. Και η οθέτηση της οδηγίας για τα εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών το Δεκέμβριο ήταν ένα πολύ καλό βήμα πρόοδου. Και αν εφαρμοστεί σωστά θα μειώσει στο ίμιση τις ε, αρνητικές συνέπειες ε, στην υγεία που έχει η ατμοσφαιρική ρήπανση. Και με συνεργασία πιστεύω ότι θα βελτιώσουμε την ποιότητα ζωή και τη διάρκεια ζωής των συμπολιτών μας. Το ίδιο και για τα χημικά. Προχωρούμε προς ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από τοξικές ουσίες, όπως ζητήσατε στο 7ο Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Δράσης. Και το πρόγραμμα βελτίωση καταλληλότητας και αποδοτικότητας του καρανιστικού πλαισίου που συνεχίζεται θα μας ε, ε, εξασφαλίσει ότι το REACH και η νομοθεσία για τα χημικά θα έχουν καλύτερα ακόμη αποτελέσματα. Σε ό,τι αφορά το νερό, προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στις ανησυχίες του κοινού για το πόσιμο είδωρ με τη νέα μας νομοθετική πρόταση. Γιατί το νερό είναι ένας πολύτιμος πόρος και θα πρέπει να τον αξιοποιήσουμε με πιο αποτελεσματικό τρόπο που θα συνάδει με την κυκλική οικονομία. Δεν έχει νόημα να χρησιμοποιούμε πόσιμο είδωρ για την άρδευση. Γι' αυτό και φέτο θα υποβάλουμε νομοθετική πρόταση για να προωθήσουμε την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λιμάτων. Και με τον Επίτροπο Φιλ Χόγκον θα προσπαθήσουμε να δείξουμε τους στενούς δεσμούς μεταξύ ύδατος και γεωργίας, ώστε και οι γεωργοί μας να υιοθετήσουν πιο βιώσιμες προσεγγίσεις κατά τη χρησιμοποίηση αυτού του πολύτιμου αγαθού. Επίσης, ένα άλλο πολύ προσφυλές θέμα στους Ευρωπαίους πολίτες είναι και η φύση. Είδα, το είδαμε αυτό στα ε, επίπεδα ενδιαφέροντος για το μέλλον των οδηγιών για τα πτηνά και τα ενδιατήματα. Και ε, το Δεκέμβριο δηλώσαμε ότι οι οδηγίες αυτές ήταν κατάλληλες ε, για τον επιδιωκόμενο στόχο και μάλιστα η δική σας ε, συμμετοχή στη διαδικασία ήταν πολύ σημαντική. Παρόλο που κρίθηκαν κατάλληλες για το σκοπό τους, οι οδηγίες για τη φύση παρόλα αυτά δεν υλοποιούν στο έπακρο του στόχους τους. Και το επισημάνατε και στο ψήφισμά σας για την ενδιάμεση αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Βιοπικιλότητα. Η αξιοποίηση του πρακτικού στο έπακρο θα εξαρτηθεί και από βελτιώσεις στην εφαρμογή των οδηγιών αυτών. Και μάλιστα έχουμε αναλάβει δέσμευση να υλοποιήσουμε αυτές τις βελτιώσεις και συνεργαζόμαστε με πολλούς άλλους επιτρόπους ε, υπό την αιγίδα του πρώτου αντιπροέδρου Φρανς Τίμερμανς προκειμένου να εκπονήσουμε ένα σχέδιο δράση για να αντιμετωπίσουμε τι ελλείψεις που ε, εντοπίστηκαν. Και μάλιστα ο δικός μου γενικός διευθυντής, ο Ντανιέλ Καγιέχα Κρέσπο, θα έρθει στην Επιτροπή σας για πιο διεξοδική ανταλλαγή απόψεων στις 21 Μαρτίου. Σε διεθνές επίπεδο επίσης έχουμε ενισχύσει τη φήμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως παγκόσμιο ηγέτη σε περιβαλλοντικά θέματα. Και μάλιστα έχουμε ενεργό συμμετοχή στην διαμόρφωση της παγκόσμιας διακυβέρνησης των ωκεανών. Και πέρυσι τον Δεκέμβριο Εγκαινιάσαμε 14 ε, δράσεις στα θέματα των κανόνων για τους ωκεανούς, ε, τα δεδομένα και την αηφόρο ανάπτυξη. Αυτό ε, αποδεικνύει και η ενεργό συμμετοχή μας στην υλοποίηση του στόχου αηφόρου ανάπτυξης, στόχο ανάπτυξης υπαριθμό 14 που προβλέπει τη συντήρηση και βιώσιμη διαχείριση των ωκεανών θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων. Και μάλιστα μια και εσείς στη Ερμόδια Επιτροπή για τη Διακυβέρνηση των Ωκεανών πιστεύω ότι θα πρέπει να εμπλακείτε πιο ενεργά και συγκεκριμένα στη συζήτηση για τους ωκεανούς και για την πολιτική μας στους ωκεανούς. Έχουμε σημειώσει αρκετή πρόοδο και στα θέματα της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών και στα θέματα των χωροκατακτητικών ειδών. Και μάλιστα έχουμε ε, πολλά θετικά αποτελέσματα σε παγκόσμιο επίπεδο χάρη στην ικανότητα συνεργασία των κρατών μελών. Τι γίνεται όμως με το μέλλον, τι άλλο μπορούμε να περιμένουμε τους επόμενους μήνες. Ε, το πλαστικό είναι ένα πολύ ευέλικτο και χρήσιμο υλικό, αλλά θα πρέπει να διαχειριστούμε καλύτερα την χρήση και διάθεσή του. Και η ευληματική μας στρατηγική για τα πλαστικά προς τα τέλη του έτους θα είναι εύχρηστη και απλή και θα έχει πολύ σημαντικά αποτελέσματα σε προβλήματα όπως τα θαλάσσια απορρίμματα. Ε, και μένουμε, μένοντα στο θέμα τη ε, κυκλικής οικονομίας, χάρη στη νέα μα στρατηγική θα έχουμε μια αναθεώρηση της συνολικής μας προσέγγισης ε, για το από πού προέρχονται τα πλαστικά, πώς θα χρησιμοποιούμε και τι θα γίνει μετά το τέλος της λειτουργίας τους. Επίσης, έχουμε αναλάβει μια πρωτοβουλία για την διασύνδεση των προϊόντων, των χημικών και των αποβλήτων στην νομοθεσία για να αντιμετωπίσουμε τα εμπόδια στην καλύτερη, στα καλύτερα ποσοστά ανακύκλωσης. Επίσης, ε, ήταν κέριος ο ρόλος μας στην ε, ανάπτυξη του θεματολογίου για το 2030 και προσυπογράψαμε και τους 17 ε, στόχους αηφορών ανάπτυξης. Η υλοποίησή τους θα ενισχύσει την υποστήριξη και την κατανόηση των Ευρωπαίων πολιτών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγκαινιάσει μία πλατφόρμα με πολλούς ενδιαφερόμενους για το ρόλο και τη συνέχιση που θα πρέπει να δοθεί στην ε, ανταλλαγή βέλτιστων των πρακτικών για την εφαρμογή των στόχων αηφόρου ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς. Οι στόχοι αηφόρου ανάπτυξης είναι και το πλαίσιο για τις τωρινές και τις μελλοντικές μας περιβαλλοντικές πολιτικές και έτσι θα εξασφαλίσουμε πραγματική και ουσιαστική πολιτική παρακολούθηση της εφαρμογής τους. Φέτος ελπίζουμε να γίνει η κύρωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της σύμβασης της Μιναμάτα προκειμένου να τεθεί σε ισχύ. Και μάλιστα θα ήθελα επευκαιρία να σας ευχαριστήσω για το έργο σας σε ό,τι αφορά το πακέτο για τον Ιδράργυρο που άνοιξε το δρόμο για την κύρωση της σύμβασης της Μιναμάτα. Έτσι ερχόμαστε πιο κοντά σε μια κοινωνία που θα είναι ασφαλέστερη, υγιέστερη και απαλλαγμένη από υδράργυρο. Ένα από τα πιο σημαντικά έργα και καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η ε, εξασφάλιση της στήριξης των υποσχέσεων των κρατών μελών, της ε, εφαρμογής δηλαδή της νομοθεσίας που από κοινού έχουν ε, εγκρίνει. Και γι' αυτό αναλαμβάνουμε δράση όταν α, διακυβεύεται το δημόσιο συμφέρον. Έτσι ενισχύουμε και το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την ποιότητα του αέρα, τα υψηλά επίπεδα διοξιδίου του άνθρακα είναι η αιτία για 70.000 πρόωρους θανάτου στην Ευρώπη το 2013. Ε, πρόκειται για αριθμό σχεδόν τριπλάσιο από τον αριθμό των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων. Ε, πρόκειται για προβλήματα που αντιμετωπίζουν τουλάχιστον 130 ευρωπαϊκές πόλεις και προβλήματα που μπορούν να αντιμετωπιστούν. Γι' αυτό λοιπόν και ξεκινήσαμε διαδικασίες ε, παραβάση κατά 12 χωρών μελών και γι' αυτό στέλνουμε και την τελική προειδοποίηση σε πέντε μεγάλες χώρες μέλη ε, ήδη από τον Ιανουάριο. Δεν μας ευχαριστεί η έναρξη τέτοιων διαδικασιών επιπαραβάση, αλλά θα πρέπει να τονίσουμε ότι είμαστε αποφασισμένοι να το κάνουμε σε περίπτωση που τα κράτη-μέλη δεν πληρούν τους στόχους και δεν εφαρμόζουν σωστά την νομοθεσία. Εγώ περιμένω την έκβαση των εργασιών της Επιτροπής εμείς για το σκάνδαλο των καυσερίων των αυτοκινήτων που θα μας οδηγήσει σε καλύτερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή ώστε να έχουμε καλύτερη ποιότητα του αέρα. Βέβαια δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε στα δικαστήρια για να εξασφαλίζουμε εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Γι' αυτό και ξεκινήσαμε τον περασμένο μήνα την αναθεώρηση τη εφαρμογή τη περιβαλλοντική νομοθεσία. Εκεί θα εντοπίσουμε του τομεί όπου τα κράτη-μέλη θα πρέπει να σημειώσουν περισσότερη πρόοδο και θα αξιοποιήσουμε τι εμπειρίε ε, με την ανταλλαγή απόψε. Έτσι θα έχουμε διετή κύκλο προσέγγισης ε, κάτι που ε, βρήκε σύμφωνος ε, τον περασμένο μήνα τους υπουργούς περιβάλλοντος όταν τους παρουσίασα τη διαδικασία για την αξιολόγηση της εφαρμογής περιβαλλοντικής μας νομοθεσίας. Γιατί πολλοί κανόνες δεν εφαρμόζονται σωστά και με συνέπεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό έχει μεγάλο κόστος για την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον. Αυτή η αξιολόγηση λοιπόν και η αναθεώρηση που θα κάνουμε είναι τίμα των προσπαθειών μας για να βελτιώσουμε την εφαρμογή ε, ώστε να έχουμε καλύτερη συμμόρφωση και καλύτερη ενημέρωση. Και το όραμά μας για το μέλλον εδράζεται στην παρουσίαση αυτών αποτελεσμάτων για τους πολίτες ό,τι αφορά το περιβάλλον με πιο ενεργό συμμετοχή και συνεργασία και όχι με παρατεταμένες ε, δικαστικές ε, διαφορές και διαμάχες. Η αποτελεσματική εφαρμογή προϋποθέτει σωστή εκτέλεση των κανόνων που εγκρίνεται ε, για να έχουμε τα αποτελέσματα που περιμέναμε με τη σχετική νομοθεσία. Σας ευχαριστώ θερμά και περιμένω τα σχόλια, τις απορίες και τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο τώρα έχουν οι βουλευτές. Πρώτα απ' όλα θα ακούσουμε τους συντονιστές ή τους αντικαθιστώντες αυτούς. Ιβο Μπέλετ, εκ μέρους του ΕΛΚΑΝ, ο πρώτος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Καλημέρα σας και σας ευχαριστούμε πολύ για την επισκόπηση όλων των σχεδίων. Ένα γενικό ερώτημα έχω. Είπατε ότι είμαστε στη μέση. Έχουμε περάσει και όλα στη μέση της θητείας. Γιορτάζουμε σύντομα τα 60 χρόνια ε, από την ίδρυση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, συνέρχονται οι αρχικοί κρατών κυβερνήσεων σήμερα στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν ε, τον τρόπο ενίσχυσης του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, Ο δικό σας ρόλο στην όλη αυτή τη διαδικασία, πώς τον αντιλαμβάνεστε. Διότι φυσικά εφαρμόζουμε τα ε, έργα και τα σχέδια. Ε, κάποια άλλα ε, θα ξεκινήσουν σύντομα. Μιλήσατε στο πακέτο Μποναφέ, θα το έλεγα εγώ το πακέτο τέλο πάντων της οικονομίας, που είπατε ότι μπορεί πολύ γρήγορα να εφαρμοστεί και το ΝΕΚ για τις, τα εθνικά νοτατόρια εκπομπών. Πώς μπορούμε να είμαστε πιο φιλόδοξοι, κύριε Επίτροπε, Βλέπουμε το πρώτο σχέδιο του εγγράφου. Θα συζητηθεί απόψε από του αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων και θα εγκριθεί στη Ρώμη. Θα οδηγήσει στην νέα διακήρυξη τη Ρώμη. Βέβαια, υπάρχει και η διάσταση τη αηφορία, τη οικονομική αηφορία και βιωσιμότητα. Πάρα πολύ σημαντικό θέμα και ίσω θα είναι και από τα βασικά σημεία της επαναδρομολόγησης του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Τα επόμενα δύο χρόνια ή δυόμιση χρόνια θα συζητούμε όμως το Brexit κατά κύριο λόγο. Και επομένως άλλη εναλλακτική από το να επαναδρομολογήσουμε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα δεν υπάρχει. Ο δικός σας ρόλος θα είναι πολύ σημαντικός. Οι συγκεκριμένες ερωτήσεις μου λοιπόν είναι οι εξής. Ποιε περαιτέρω πρωτοβουλίε συγκεκριμένε πέραν του πλαστικού και των θεμάτων που ήδη έχουν δρομολογηθεί μπορούν να αναλυφθούν, θα μπορούμε να σχεδιάσουμε νέε πρωτοβουλίε, να εφαρμόσουμε νέε πρωτοβουλίε για αυτά τα επόμενα 2-2,5 χρόνια και σε ό,τι αφορά την Ευρώπη των πολλαπλών ταχυτήτων, ενισχυμένη συνεργασία μιλάμε. Ε, αλλά σε περί, επίπεδο 27-28 δεν ξέρω αν αυτό είναι δυνατόν. Τι άποψη έχετε για την Ευρώπη πολλαπλών ε, ταχυτήτων και στους τομείς χαρτοφυλακίου σας. Θα υπάρχουν κάποια κράτη που ενδεχομένω θα θέλουν να προχωρήσουν περισσότερο. Η δική σα χώρα προεδρεύει τη Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το εξάμεινο είσαστε λοιπόν σε μια ιδιαίτερη θέση. Εμείς είμαστε στο σταυροδρόμι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς μπορούμε λοιπόν, τώρα που θέλουμε, να το αξιοποιήσουμε αυτό το δυναμικό ε, στις οικονομίες μας, ε, γιατί μίλησατε κι εσείς για ευημερία των πολιτών. Προς το σκοπό αυτό λοιπόν, πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε και να είμαστε πιο φιλόδοξοι τα επόμενα δυόμιση χρόνια. Ευχαριστώ. If it's okay for you. It's okay. Okay. So, Κύριε Μπέλετ, σας ευχαριστώ πολύ για το πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Όπως είπατε, είμαστε στη μέση της ε, θητείας και έχουν περάσει 60 χρόνια από την ε, έναρξη αυτού του οικοδομήματος, από την ίδρυση που θα ε, γιορτάσουμε στη Ρώμη που δεν θα τη γιορτάζαμε αν δεν είχαμε πολλά πλεονεκτήματα και ωφέλη ήδη. Αν έχει κρατήσει αυτή η υπόθεση 60 χρόνια, αν δεν μας είχε δώσει όμως κάποιο όφελος, δεν τη γιορτάζαμε. Το ότι τη γιορτάζουμε σημαίνει ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε τα ωφέλη που έχουν αποκομίσει τα κρατημέλη και οι πολίτες, ε, όπως είπατε και εσείς, οι συμπολίτες μας. Πολλά κάναμε, Πολύ έχουμε προχωρήσει σε ό,τι αφορά την ποιότητα του αέρα, τη γλυκή οικονομία, τη βιοπικιλότητα, τη φύση κτλ. Φυσικά πολλά ακόμα από να γίνουν, αλλά αν δείτε ποια ήταν η δική μας εντολή, θα δείτε ότι σχεδόν όλες οι ιδέες που είχαμε, χάρη σε εσά και τους συναδέλφους μας στο Συμβούλιο, από νομοθετικής πλευράς, σχεδόν έχουμε ολοκληρώσει το θεματολόγιό μας. Γιατί λέω ε, νομοθετικά μιλώντας. Διότι, αν δούμε προς το μέλλον, πρέπει πλέον να εστιάσουμε στο σημαντικότερο, που είναι η εφαρμογή, η υλοποίηση. Έχει νόημα να συσσωρεύουμε το ένα νομοθέτημα μετά το άλλο, εάν αυτά τα νομοθετήματα δεν εφαρμόζονται. Επιλέγουμε λοιπόν είτε να αυξήσουμε τα νομοθετήματα, είτε να φροντίσουμε τα υφιστάμενα όχι απλά να εφαρμόζονται, αλλά να εφαρμόζονται πλήρως. Εγώ εκεί θα εστιάσω και στο μέλλον, στον τομέα δηλαδή της εφαρμογής, της υλοποίησης και νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι, όπως είπατε και εσείς. Και νομίζω ότι σε ό,τι αφορά το επίπεδο φιλοδοξίας, ε, η Κομισιόν είναι πολύ πιο κοντά το Κοινοβούλιο, σε σχέση με τα άλλα θεσμικά όργανα που φυσικά βέβαια πρέπει να καταλήξει και στο τελικό συμβιβασμό. Υπάρχει όμως και μια άλλη είδους φιλοδοξία που δεν αφορά μόνο τη στοχοθέτηση ή τα επίπεδα των προτύπων που θέλουμε να πετύχουμε. Φιλοδοξία είναι στον καλύτερη περίπτωση να φροντίσουμε να υπάρχει και εφαρμογή, κύριε Μπέλετ. Και ναι, φυσικά είπατε ότι πρέπει να είμαστε φιλοδοξοί και στους στόχους, αλλά και στην εφαρμογή τουλάχιστον, που είναι και ίσως και πιο σημαντικό, αν θέλουμε να έχουμε αυτά αποτελέσματα. Σε ό,τι αφορά την Ευρώπη των πολλαπλών ταχυτήτων, αυτή είναι μια επιλογή. Περιλαμβάνεται στη Λευκή Βίβλο προσυζήτηση και νομίζω ότι θα είναι ένα από τα ζητήματα που θα συζητηθούν περισσότερο στο άμεσο μέλλον. Και από ό,τι βλέπω, ενδεχομένως θα υπάρξουν διαφορετικές τάσεις. Ε, κάποια κράτη-μέλη μπορεί να θέλουν να προχωρήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Ίσως για διαφορετικά, για διαφορετικούς λόγους, λόγω διαφορετικών συμφερόντων το καθένα. Έχει τα υπέρ και τα κατά του αυτό. Γιατί όταν συζητούμε, όταν μιλούμε για ευρωπαϊκό οικοδόμημα συνήθω, δεν μας απασχολεί το ποιος θα φτάσει πρώτος, αλλά όλοι πρέπει να φτάσουμε Είμαστε 28, θα γίνουμε 27 μάλλον, πολύ σύντομα. Αλλά δεν κάνουμε αγορά ταχύτητα. Ποιο θα φτάσει στον τερματισμό. Και 27 πρέπει να τερματίσουμε. Άρα, όταν μιλάμε για μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων, εγώ προσωπικά δεν θα ήμουν υπέρ. Αν αυτό σημαίνει εγώ τα κατάφερα, τερμάτισα, έβαλα γκολ, δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι υπόλοιποι. Θα πρέπει να αλληλοϊποστηριζόμαστε. Έτσι υπάρχουν κάποιοι που πηγαίνουν πιο γρήγορα και συμφωνώ ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει πρόβλημα όταν κάποιο θέλει να προχωρήσει πιο γρήγορα. Έχουμε τα κράτη-μέλη που πηγαίνουν με 28 διαφορετικές ταχύτητες σήμερα. Το θέμα είναι όμω ότι πηγαίνουν προς την ίδια κατεύθυνση και ασκηνούνται με διαφορετικούς ρυθμού. Η καταστροφή θα ήταν να μην πήγαιναν όχι μόνο με διαφορετική ταχύτητα, αλλά και σε διαφορετικές κατευθύνσεις τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, ο κύριο Πάβελ Πότσο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αλλά και εσά Επίτροπε, που ήρθατε και για τα όσα μας εξηγήσατε για τις ε, απαντήσεις σας ναι, για τα φυτοφάρμακα για τα λοιπάσματα τέλος πάντων θέλουμε και εμείς να γίνουν αυτές οι περικοπές σε κάδμιο και έτσι να εκτίθενται λιγότερο οι Ευρωπαίοι και να προστατεύουμε από τις τοξικές αυτές ουσίες τους Ευρωπαίους. Είναι, δεν είναι στο γραπτοφυλάκιό σας. Μπράβο που έχετε τόσο ξεκάθαρε θέσει. Τώρα θα ήθελα να σας ρωτήσω για κάτι διαφορετικό. Κάτι το οποίο βρίσκεται ψηλά στο θέμα τη Γενικής Διεύθυνση για την Υγεία. Είναι ένα από τα πολλά προβλήματα για τη δημόσια υγεία. Για τις τοξικές ουσίες που υπάρχουν στο περιβάλλον και κυρίως στη θάλασσα και, μπορούν να σκοτώσουν πολλά ήδη. Πολύ σωστά τα όσα κάνατε για την οδηγία που αφορά τους βιότοπους και τα πτηνά όπως ήθελε και κοινή γνώμη, συνεχίσατε την πορεία αυτών των οδηγιών και πέστε μας τι θέλει να κάνει τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτή την οδηγία που είναι τόσο σημαντική ε, γιατί όσον αφορά την προστασία και καλομεταχείριση των ζώων είναι κάτι που ενδιαφέρει πολλούς εμπλεκόμενους. Στις 2 Μαρτίου έγινε η συνάντηση με τους Κινέζους. Τι θα γίνει το 2017 στα πλαίσια της πλατφόρμας των σχέσεων με την Κίνα. Θα σε ευχαριστώ κύριε Πότσο και πρώτα πρώτα να σας πω τι γίνεται με αυτούς τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Όπως ξέρετε ασχολούμεθα πολύ με το θέμα και με μεγάλη προσοχή προχωρούμε. Οπότε θα προσπαθήσουμε να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση. Για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τους διαταράκτες. Τώρα ε, μας είπατε για τα λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα και για το πρόβλημα του καδμίου. Όπως γνωρίζετε, είναι η περιεκτικότητα των τροφίμων σε κάδμιο είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα της υγείας. Έχουμε από τα φωσφορούχα μόλυνση των γεών που χρησιμοποιούνται για γεωργία. Και εμείς είμαστε υπέρ του να αναθεωρηθεί ο σχετικός κανονισμός για τα φυτοφάρμακα και να μειωθεί η περιεκτικότητα σε κάδμιο. Άλλωστε εκκρεμεί το θέμα πάνω από μια δεκαετία. Ήρθε η ώρα να κάνουμε κάτι και να έχουμε υλικά που δεν είναι τοξικά και να επιδέχονται και ανακύκλωση γιατί το θέμα δεν είναι τι, γίνεται ε, με τη μία χρήση, την εφάπαξ χρήση το θέμα είναι τι γίνεται συνεχώς άρα χρειάζεται ανακύκλωση και εν προκειμένου τέτοια προσέγγιση έχουμε από οπτικής γωνίας κυκλικής οικονομίας δεν θέλουμε τα βιοαπόβλητα να συνεχίσουν να ανακυκλώνονται και να υπάρχει σορευόμενη μόλυνση και ρήπανση. Νομίζω είναι ρεαλιστικές οι προτάσεις μας. Και νομίζω ότι μπορείτε και εσείς να προωθήσετε ε, τις προτάσεις σας, ακόμα και πριν αποφασίσει επόμενο τομέα στο Συμβούλιο. Τώρα, όσον αφορά αυτό τον έλεγχο επιδόσεων του, για τα νομοθετήματα για τη φύση. Αυτό το fitness check οι σχετικές οδηγίες καλώς τα πήγανε απ' την άλλη όμως δυστυχώς ακόμα και αν είναι δόκιμες για επίρρευση του σκοπού τους οι οδηγίες δεν θα πιάσουν το από εκτός εάν αρχίσουμε να τις εφαρμόζουμε με σοβαρό τρόπο Είχαμε πέρσι την έκθεση για την κατάσταση των πραγμάτων σχετικά με την φύση και λοιπά, τη στρατηγική για την βιοπικιλότητα και όλες αυτές οι μελέτες και εκθέσεις έλεγαν ότι ε, οι στόχοι μας για τη βιοπικιλότητα και για τη φύση δεν θα επιτευχθούν. Τούτο δε μας προβληματίζει η βιοπικιλότητα συνεχίζει να επιδεινώνεται. Δεν ξέρω, ε, έχουμε ε, μια εξής τελευταίας ε, τετραετίας. Δεν πρόκειται αυτό να φρενάρει και να αναστραφεί το κλίμα σε τέσσερις μήνες, αλλά τουλάχιστον κάτι να αλλάξει και όπως γνωρίζετε. Μαζί σας και άλλους συναδέλφους είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρξει σχέδιο δράσης για το πώς οι οδηγίες για τη φύση θα υλοποιηθούν καλύτερα. Και αυτό το πρόγραμμα δράσης πρόκειται τις αμέσως επόμενες εβδομάδες να ξεκινήσει επί τη βάση των επιδόσεων των ε, αποτελεσμάτων των διαβουλεύσεων αλλά και των εκθέσεων που έχουν γίνει στο μήκο κύματος των όσων εσείς έχετε ζητήσει για βελτιώσεις στην υλοποίηση των νομοθετημάτων. Τώρα, όσον αφορά τις επαφές με την Κίνα για τους ωκεανούς, θα ήθελα να σας ζητήσω το εξής. Η δική σας επιτροπή είναι κυρίως αρμόδια για τους ωκεανούς και γνωρίζω ότι οι Πορτογάλοι συνάδελφοι εδώ ασχολούνται με το θέμα. Ξέρω ότι έχετε αναπτύξει. Πού είστε. Α, εδώ είναι, εδώ είναι. Εδώ είναι. δεν έχω τα γυαλιά μου, κυρία μου, γι' αυτό δεν σας είδα. Ξέρω ότι έχετε αναπτύξει τα δραστηριότητα, αλλά νομίζω ότι αν συναντηθούμε ε, ε, επανειλημμένα θα υπάρξει και ενημέρωση, γιατί το θεματολόγιο του ωκεανού δεν είναι κάτι που αφορά μόνο την Ευρώπη. ή ωκεανοί είναι το περιβάλλον, το οποίο δεν διαιρείται σε κινέζικο, αμερικάνικο, ευρωπαϊκό. Είναι παγκόσμιο το περιβάλλον οι ωκεανοί αφορούν όλη την υδρόγειο. Και τα προβλήματα επομένως είναι παγκόσμια και επιδέχονται άρα παγκόσμιες λύσεις που θα έρθουν με παγκόσμια δράση. Πέρσι είχαμε εκδώσει και δημοσιοποιήσει κάποια ανακοίνωση όσον την διακυβέρνηση ε, της πολιτικής των ωκεανών γύρω από τρεις άξονες πρώτα-πρώτα να αναβαθμίσουμε το σημερινό νομοθετικό πλαίσιο. Έχουμε ε, του τους κανόνες ον UNCLOS πολύ αλλά υπάρχουν κάποια κενά στο νόμο για την διακυβέρνηση, για την βιοπικιλότητα, πέραν ε, των ε, εθνικών συνόρων και δικαιοδοσιών. Δεύτερος άξονα είναι το πώς θα μειώσουμε ή πώς θα σταματήσουμε την ε, βλαπτική δράση των ανθρώπων για τους ωκεανούς μας. Μεγάλο πρόβλημα. Είναι αυτά τα θαλάσσια απόβλητα. Φυσικά τα θαλάσσια απόβλητα προέρχονται από την ξηρά και λοιπόν του ωκεανού. Οπότε θα πρέπει αυτού του είδου η ανθρώπινη πίεση να αρθεί, να μειωθεί. Και τρίτο άξονα είναι ότι θα πρέπει να αποκτήσουμε καλύτερη γνώση των ωκεανών μα. Συχνά λέμε ότι ο άνθρωπος πήγε από τη γη στο διάστημα μέσω του ωκεανού. Βεβαίω, έχουμε επενδύσει πολλά, έχουμε ξοδέψει πολύ χρήμα για έρευνα στην Αρκτική, στους ωκεανούς, παντού. Άρα σε αυτόν τον ε, τρίτο άξονα θέλουμε να εντάξουμε μεγαλύτερη πρικοδότηση, μεγαλύτερες δαπάνες για να μάθουμε τους ωκεανού μας. Και έχουμε διεξαγάγει επαφές και συζητήσεις με όλους, με ΙΠΑ, με Κίνα, με τις χώρες της Αφρικής και με την Κίνα. Πολύ ενδιαφέρουσαν οι επαφές. Η πρώτη μου συνάντηση έγινε σχεδόν πριν από δύο χρόνια. Και μίλησαμε την ίδια γλώσσα και ανταλλάξαμε πληροφορίες, εμπειρίες και διαπιστώσαμε ότι ενδιαφέρει πολύ το θέμα τους Κινέζους. Φέτος δε έχουμε το γαλάζιο έτος που αφορά Κίνα και Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχουμε διασκέψεις πολλές για τους ωκεανούς φέτος. Την προηγούμενη, τον προηγούμενο μήνα στην Ινδονησία έγινε η διάσκεψη του Economist και η Γενική Διεύθυνση 14 θα συμμετάσχει στη διάσκεψη του ΟΗΕ που θα γίνει στη Νέα Υόρκη. Και η Σουηδία επίσης ε, με τα νησιά Φίτζη υποστηρίζει αυτή την διάσκεψη του ΟΗΕ. Και έχουμε επίσης και στην Μάλτα. 5 και 6 Οκτωβρίου μία διάσκεψη. Τέταρτη διάσκεψη. πρώτη έγινε ο Άσμα, μετά στη Χιλή, τρίτη στην Ουάσιγκτον και η τέταρτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη Μάλτα. Η πέμπτη διάσκεψη θα γίνει στην Ινδονησία. Στη συνέχεια δε, η επόμενη στην Νορβηγία. Σας ευχαριστούμε λέει η Πρόεδρος. Έχουμε πολλούς ομιλητές. Τώρα από ε, ομαδοποιήσουμε κάποιες ερωτήσεις. Ο κύριος Ντεμές Μάκερ τώρα από την πολιτική ομάδα ECR να σας τα πω στα Ολλανδικά. Καλώς ορίσατε κύριε Επίτροπε. Εισαγωγικά μας είπατε ότι η Επιτροπή περί τα τέλη της Άνοιξης αποφάσισε να μην πάψει η ισχύ της οδηγίας για τους βιότοπους και τα πτηνά. Μπράβο. Χαιρόμαστε γι' αυτό και εγώ και άλλοι συνάδελφοι που θεωρούμε ότι αυτό ήταν μια ορθή επιλογή. Γιατί έχουμε μια σειρά μελετών που δείχνουν ότι δεν υπάρχει κάτι στραβό με αυτή την οδηγία. Το πρόβλημα είναι η υλοποίηση, η εφαρμογή της. Εδώ θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας. Ε, αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να στείλουμε σε όλους αυτούς τους Ευρωπαίους που κάνουν ό,τι μπορούν κάθε μέρα για να προστατευτεί η βιοπικιλότητα. Μας είπατε επίση για το πρόγραμμά σας, το πρόγραμμα δράσης που θα ξεκινήσει μετά το τέλος της Άνοιξης, αλλά για πέστε μας δύο λόγια για το περιεχόμενο αυτού του προγράμματος δράσης που δεν μας εξηγήσατε. Και αυτό είχε τονιστεί στην έκθεση του Φεβρουαρίου ότι η προστασία της βιοποικιλότητας αλλά και άλλες σχετικές πολιτικές είναι πάρα πολύ σημαντικές και για ε, την δασική πολιτική αλλά και για τη γεωργία. Διάβεστε μας πώς συνεργάζεστε με άλλους συναδέλφους σας ούτως ώστε αυτό το πρόγραμμα δράσης που εξαγγείλατε πρόκειται να βοηθήσει για να υπάρξει αυτού του είδους ολοκλήρωση αυτού του είδους αλληλεπίδραση των διαφορετικών τομέων γιατί ακριβώς η βιοπικιλότητα ε, απαιτεί πολυτομιακή προσπάθεια. Δεν πέστε μας το πώς θα γίνουν αυτά. Τελευταία με ερώτηση. Τι γίνεται με το εαρινό κυνήγι όσον αφορά τα μεταναστευτικά πτηνά. Μέσω της ε, σχετικής οδηγίας θα θεσπίσετε τα κατάλληλα μέτρα. Έχετε πει ότι θα το κάνετε. Θέλουμε να δούμε να αναλαμβάνετε δράση. Που είναι σημαντικό αυτό για την ε, αξιοπιστία μας έναντι των Ευρωπαίων. Ευχαριστώ κύριο της άλλης κύριο Γκερμπράντη. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω και τον Επιτροπό που είναι εδώ για μια ακόμη φορά μαζί μας. Την ε, προηγούμενη φορά όταν σας συναντήσαμε, συζητήσαμε και την ενδιάμεση αναθεώρηση της στρατηγικής για τη βιοπικιλότητα και εγώ σας περιέγραψα ε, με αδρές γραμμές ε, την ε, κατάσταση που περίμενα να επακολουθήσει μετά την δημοσιοποίηση της κατάστασης της φύσης. Είναι κατεπήγον το θέμα. Ξέρω ότι τότε ελληνική θητεία του Προέδρου της ε, Κομισιόν. Ήμασταν πολύ μακριά όμως από την επίτευξη των στόχων περιβιοπικιλότητας και ακόμα χειρότερα ήταν ε, πολύ χαμηλότερα τα ποσοστά όλων των δικτών ε, από ό,τι θα έπρεπε. Μειώνονταν για τη βιοπικιλότητα. Τι έγινε τελικά. επίθεση σε βάρο τη οδηγία για την προστασία των πτηνών και από το ίδιο το πολιτικό γραφείο του Προέδρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διότι αν υπάρχει ένας υπεύθυνος ε, για την καθυστέρηση της όλης διαδικασίας για την ε, προστασία της οδηγίας αυτής και την υποστήριξη της οδηγίας για την προστασία των ποινών, δυστυχώς πρέπει να πω ότι αυτός είναι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δέχεστε λοιπόν ε, να ακολουθήσετε μια άκρος επιθετική προσέγγιση προκειμένου να βελτιώσετε τις ε, πολιτικές ε, και την εφαρμογή σε ό,τι αφορά τη βιοπικιλότητα, διότι μετά τη δημοσίευση της κατάστασης της Free State of Nature τα πράγματα ε, πήγαν αντίστροφα, έγινε το αντίστροφο αυτό που θα έπρεπε. Ίσως αυτή η εικόνα που είδαμε χθε στη Μάλτα με την καταστροφή του μπλε παραθύρου είναι μια εικόνα για το τι συμβαίνει τώρα. Τι θα κάνετε τώρα, πέραν της δημοσιοποίησης του σχέδιου δράσης, γιατί γνωρίζουμε ότι δεν επαρκεί αυτό. Η γεωργία. Γνωρίζουμε ότι είναι ένας από τους βασικούς λόγους ε, για την απώλεια βιοπικιλότητας. Χρειαζόμαστε τους ε, αγρότες, αλλά αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να τους εισπυρώσουμε πίσω από τον ίδιο στόχο. Στην Επιτροπή Λεκτού Προπολογισμού πριν από κάποιες εβδομάδες ε, ρώτησα τον ε, Τόπο Χόγκαν να μου πει τι περιμένει αυτό τις επόμενες εβδομάδες και μήνες και μου είπε περιμένετε ε, να έρθει η επόμενη κοινή γεωργική πολιτική, δηλαδή μετά το 2021. Θα έχει λήξει προθεσμία όμως τη στρατηγική για τη βιοπικιλότητα. Πώς θα πείσετε λοιπόν τους συναντέλφου σας, τι θα κάνετε για να του πείσετε ότι είναι απαραίτητο να αναλάβουν δράση. Ένα άλλο παράδειγμα για να δείτε πού βρισκόμαστε. Με το δάσος της Βιλοβίτσας στην Πολωνία. Ξέρετε τι έγινε. Πήρατε δράση, αναλάβατε δράση και θέλω να σας συγχαρώ για αυτό. Τι γίνεται όμως, συνεχίζεται η άσκηση πιέσεων. συνεχίζεται συγγνώμη, η παράνομη και η ζημιά είναι ήδη ανεπανόρθωτη. Εγώ νομίζω ότι χρειάζεται μια στρατηγική. Διαφορετική ίσως από αυτή που έχετε ακολουθήσει μέχρι τώρα. Υπάρχει ένα σχέδιο έκτατης ανάγκης. Ευχαριστώ. Θέλετε να απαντήσετε. Έχω και άλλους δύο συντονιστές. γιατί θα να καθυστερήσουμε. Πού είναι Γκουε, Μπόλαν. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ και τον Επιτρόπο που ήρθε εδώ να μας δώσει τη δυνατότητα να θέσουμε ερωτήσει. Έχω ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα για το νερό. Ρωτώ την Κομισιόν γιατί, κύριε Επίτροπε, δεν λαμβάνετε υπόψη τις δημοκρατικές επιθυμίες ε, των ε, συμπολιτών σας. Ε, το Μάιο του Είχαμε 1,8 εκατομμύρια υπογραφές και ζητήθηκε από την Κομισιόν να εγγυηθείτε την, ε, την ε, υδροδότηση της υπηρεσίας για της αποχέτευσης, ε, να μην υπάρξει απελευθέρωση, τον Οκτώβριο του 2014 η Αρμόδια Επιτροπή εδώ ενέκρινε μια έκθεση υπέρ της πολιτών. Το 2015 το Σεπτέμβριο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ενστενίστηκε τις δημοκρατικές επιθυμίες των πολιτών. Έκτοτε έχουμε κοφαντική σιγή από πλευρά της Κομισιόν. Δεν έχει δοθεί καμία όθηση στην αντιμετώπιση ε, και στην ανταπόκριση σε αυτό το αίτημα των πολιτών ε, και του Κοινοβουλίου μας και ιδίως για την περίπτωση της Ιρλανδίας και το νερό. Είναι τόσο αποτελεσματική μονάδα που έχει δημοσιοποιήσει μία γραπτή ε, ερώτηση, απάντηση μάλλον σε ένα δημοσιογράφο. Και χρειάστηκε καταγγελία στον Ευρωπαίο Διανοσολαβητή. Πότε θα αρχίσετε να σέβεστε τη δημοκρατία να ανταποκριθείτε ε, σε αυτό το έτοιμο και το κίνημα των πολιτών για το νερό. Θα είστε ουδέτεροι σε σχέση με το νερό ως ανθρώπινο δικαίωμα και το πώς ε, θα το χειρίζεται το θέμα του νερού το κάθε κράτος μέλος. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Έκχατ είναι ο τελευταίος από το κατάλογο των συντονιστών που λαμβάνει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον Επίτροπο που ήρθε στη συνεδρίαση. Όντως, παρακολουθήσατε και εφαρμόσετε κατά γράμμα την επιστολή ανάθεση καθηκόντων ε, που σας έδωσε ο κύριος Γιουνκέρ κατά την άρξη θητείας. Βέβαια, το μόνο που αφορούσε ε, η επιστολή ήταν η καλύτερη νομοθεσία για το περιβάλλον, δηλαδή η εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας ε, που είχε ήδη εγκριθεί στα πλαίσια του προκατόχου σας και μόνο η οδηγία για, τη, για τα ενδιατήματα και τα πτηνά ε, αναφερόταν στην επιστολή. Οπότε ήταν σχετικά εύκολο το καθήκον σας. Ε. Οπότε δεν είχατε και πολλά. Ε, βέβαια μετά τις εξελίξεις ε, ε, που δεν ε, ήσταν πιο ε, ενεργός και δεν ε, κάνετε περισσότερες δηλώσεις. Καταρχήν, συνεχίζεται η, συζήτηση για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και ουσιαστικά ε, αλλοιώθηκαν τα μέτρα του πρασινίσματος στην ΚΑΠ ε, είναι σαν να λέτε και τώρα θα ελέγξουμε ποιοι δεν κάνουν, δεν εφαρμόζουν σωστά την νομοθεσία. Ο προκάτοχός σας ε, ήταν πολύ πιο δραστήριο ό,τι αφορά το πρασίνισμα τη ΚΑΠ. Ε, με εσά δεν είμαι και πολύ σίγουρο ότι το λαμβάνετε σοβαρά υπόψη. Και οι νέε προτάσει για την ΚΑΠ ε, δεν έχουν καν υποβληθεί. Και αυτό είναι ε, θεμελιώδου σημασία αν θέλουμε να διαφυλάξουμε τη βιοποικιλότητα. Θα ήθελα μια πολύ πιο δραστήρια Γενική Διεύθυνση περιβάλλοντο. Τα τελευταία δυόμιση χρόνια ήταν σχετικά δρανή η Γενική Διεύθυνση περιβάλλοντο. Επίση, δεν αναφερθήκατε καν στο Dieselgate, στο σκάνδαλο με τα καυσαέρια δεν το προσέξατε, δεν, ε, δεν αντιληφθήκατε ότι συνέβη κάτι τέτοιο και δεν ε, αντιληφθήκατε ότι ήδη δημοσίευσε η εμείς την έκθεσή της που καταδικάζει και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταξύ άλλων. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, λοιπόν, θεωρώ ότι πρέπει να λάβει πολύ σοβαρά υπόψη την έκθεση της εμείς. Ξέρουμε ότι δρομολογούνται κάποιες βελτιώσεις, αλλά έχουμε, ε, εξακολουθούμε να έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα πολύ ρηπογόνα αυτοκίνητα εξακολουθούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Θέλουμε περιβαλλοντικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις που αυτή τη στιγμή στερούν. Ο προκάτοχός σας είχε ήδη ετοιμάσει πρόταση για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις, αλλά αρχιοθετήθηκε εξαιτία αυτή τη περιβόητη καλύτερη νομοθεσία, γιατί δεν θεωρήθηκε σημαντικό. Αυτό όμω που έδειξε το Dieselgate είναι ότι πραγματικά είναι σοβαρό το θέμα, γιατί αφορά την υγεία των συμπολιτών μα. Γιατί λοιπόν δεν μα είπατε κουβέντα για το θέμα αυτό, ότι θα επαναφέρετε την πρόταση του προκατόχου σα. Να δώσουμε μία μάχη, γιατί πραγματικά διακυβεύεται το περιβάλλον και θέλω έναν επίτροπο που θα δώσει μάχη για το συμφέρον και την υγεία των πολιτών μας. Ευχαριστώ. και η κυρία Μαγκίνες. Ε, ε, θα ήθελα να ζήσω την επικιά της και να της δώσω τώρα το λόγο γιατί πρέπει να φύγει για άλλη συνεδρία. Σε ευχαριστώ αγαπητή κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους συναδέλφους που με επιτρέπουν να λάβω τώρα το λόγο. Ευχαριστώ τον Επιτροπό για την παρουσίασή του και για την ε, επιμέρους ενημέρωση για θέματα. Εγώ θα συνεχίσω αυτά που είπε ο προλαλής σας για την γεωργία. Γιατί ε, με ενοχλεί αυτό το ψευδορήγμα μεταξύ περιβαλλοντολόγων και γεωργών. Γιατί όπως είπε και ο κύριος Δεμεσμέκερ, θέλουμε γεωργούς που θα έχουν θετική δράση και θα παράγουν τρόφιμα αλλά και θα προστατεύουν το περιβάλλον. Δεν ε, συμφώνω με αυτή την αντιπαράθεση. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να γεφυρώσει αυτό το χάσμα μεταξύ περιβαλλοντολόγων, οικολόγων και γεωργών. Αν δεν τα καταφέρουμε, θα έχουμε αποτύχει και στου δύο κλάδου, και στη γεωργία και στο περιβάλλον έχω επαφή με νέους γεωργούς που τους λέω εσείς θα πρέπει να είστε και οι περιβαλλοντολόγοι και οι γεωργοί ταυτόχρονα. Και στη συνεργασία με μη κυβερνητικέ οργανώσει θα πρέπει να επιταχύνουμε τα πράγματα. Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Γιατί ε, κνευρίζονται και απογοητεύονται και οι περιβαλλοντολόγοι και οι γεωργοί. Και υπάρχουν ε, τεράστια χάσματα, τεράστια ρήγματα και αντιπαραθέσει μεταξύ του που δεν βοηθούν κανέναν. Επίση ε, αλία χαμηλού αντικτύπου, θα το ξέρετε φαντάζομαι, και την ενδιαφέρουσα ταινία για μια παλήρια καμπή για την ανθρώπινη ζωή. Και αυτό το θέμα μας είναι πολύ ενδιαφέρον και προσφυλές. Γιατί μερικοί αντιδρούν κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί κρίνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξυπηρετεί μόνο τους ε, ισχυρούς. Είτε αυτοί είναι αλλοί, είτε επιχειρηματίες, είτε οτιδήποτε. Προσοχή λοιπόν, να στηρίξουμε και αυτού που ασκούν αλληλεία χαμηλού αντικτύπου. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τι ανησυχίε του, όπω αναφέρονται σε αυτό το έντυπο και στη σχετική ταινία. Λυπούμε που και σα ζητώ και το προτέρω συγγνώμη γιατί θα πρέπει να φύγω, αλλά θα αφήσω τη βοηθό μου για να ακούσει τι απαντήσει σα. Ευχαριστώ, πλειάδα ερωτήσεων και θα ακολουθήσουν και άλλε στη συνέχεια, αλλά α ακούσουμε τώρα τον Επίτροπο για να μα απαντήσει σε αυτά που έθεσαν μέχρι τώρα οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να ομαδοποιήσω τα ερωτήματα ώστε να απαντήσω από κοινού. Σε ό,τι αφορά την οδηγία για τα ενδιατήματα, νομίζω ότι η στόχοι του σχεδίου δράσης Φυσικά και πρώτα απ' όλα θα πρέπει να, λαμβάνουν, να λάβουν υπόψη τα σχόλια που έχουμε λάβει και θα πρέπει να αντιμετωπίσουν ε, τα βασικά αιτία τη υποβάθμισης τη βιοπικιλότητα. όπω αναφέρουν περισσότερε εκθέσει Σε όλε τι εκθέσει, η γεωργία είναι πάντοτε στην πρώτη θέση, είναι η, η πρώτη αιτία, αλλά θα επανέλθω σε αυτό. Το σχέδιο δράσης θα αντιμετωπίσει φυσικά ε, τη συνεκτικότητα με τους κοινωνικο-οικονομικούς στόχους, θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει το πλήρες δυναμικό για να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε υγιή οικοσυστήματα, ακόμα και με την συμμετοχή και των οικονομικών κλάδων. Γιατί δεν μπορείς πλέον να ε, έχεις αυτό το χάσμα, τη διαίρεση μεταξύ περιβάλλοντος, αγροτών και οικονομικών περιβαλλοντικών τομέων. Αυτό που λέμε είναι ότι πρόκειται για μια τεράστια περιβαλλοντική πρόκληση, η οποία όμως ενέχει και οικονομικές ευκαιρίες. Ό,τι αφορά τη συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων, οφείλω να πω ότι τα κράτη με ελληνική όλοι, οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν ε, συμμετάσχει ήδη από τη φάση της διαδικασίας διαβούλευσης, από την αρχή της όλης διαδικασίας συμμετέχουν και ενεργά και ιδίω στη φάση της ε, προετοιμασίας. Και όλοι όσοι ενεργά συμμετείχαν στις διαβουλεύσεις θα συμμετάσχουν το ίδιο ενεργά και στην εφαρμογή. Πρέπει να πιέσουμε τα κρατημέλη της εμπλεκομένης φορείς ώστε να εφαρμόσουν το σχέδιο δράσης το οποίο θα συμφωνήσουμε από κοινού. Αυτό το σχέδιο δράσης θα το καταρτήσουν ε, μια ομάδα από επιτρόπους με επικεφαλής τον πρώτο αντιπρόεδρο, τον κύριο Τίμερμαντ. Στο Συμβούλιο λογικά θα έχει εγκρίνει τα ε, συμπεράσματά του κάποια στιγμή τον Ιούνιο. Οπότε το Κοινοβούλιο ρωτώ αν θα έχει κάποιο ψήφισμα για αυτό το σχέδιο δράσης. Φυσικά εμείς θα δούμε σε αυτό το σχέδιο δράσης και άλλα θέματα τα οποία ίσως δεν είχαν εξεταστεί επαρκώς και καλυφθεί επαρκώς από τις ε, στάμενες ε, οδηγίες, ε, πράσινες υποδομές, επικονίαση και να δούμε και εκτός των περιοχών Natura 2000 τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό το σχέδιο δράσης γιατί υπάρχει βιοπικιλότητα και εκτός του δικτύου Natura 2000. Και επειδή μιλούμε για την ε, Natura 2000 και τις περιοχές, μιλάμε για προστατευόμενες περιοχές στην ξηρά. Έχουμε φτάσει γύρω στο 20% της ε, χερσίας μάζας. Όταν μιλάμε όμως για θαλάσσιες ε, προστατευόμενες περιοχές, πρέπει να καταλάβουμε ότι οι ωκεανοί μας εχουν πανω πάνω από 65-70% του της βιοπικελότητας του πλανήτη. Άρα όταν μιλάμε για βιοπικιλότητα μην εστιάζουμε μόνο στην γη, στην ξηρά, αλλά και στη θάλασσα, στους ωκεανούς. Για τις περιοχές λοιπόν Natura 2000, στο σχέδιο ΔΑΣ και θέλω να το τονίσω, θεωρούμε ότι αρκεί να ταυτοποιήσουμε αυτές τις περιοχές. Το 20% είναι είπα και πριν. Όμως, διαχειριζόμαστε και διαχειριζόμαστε καλά αυτές τις περιοχές. Και σε ποιο ποσοστό. Η απάντηση είναι γύρω στο 50%. Δεν μιλώ καν για το 20% των περιοχών του Natura 2000, αλλά για το 10% που έχει αναγνωριστεί και που είναι υποδιαχείριση. Έρχομαι τώρα στη γεωργία. Πράγματι σε όλες τις εκθέσεις που σας ανέφερα, κατάσταση περιβάλλοντος της φύσης, Ενδιάμεσα αναθεώρηση, η Γεωργία βρίσκεται πάντοτε στην πρώτη θέση μεταξύ των αιτιών. Όπως είπε η κυρία Μακίνης. Λύσεις χρειάζονται. Ο στόχος μας για να τις ε, εξεύρουμε αυτές τις λύσεις δεν είναι να κατηγορούμε κανέναν. Οι αγρότες είναι και πρέπει να είναι τμήμα της λύσης μιλάμε για επιβλαβή λιπάσματα. Οι επιστήμονες ε, τα παρασκεύασαν, όχι αγρότες, και τα περισσότερα λιπάσματα τα έχουμε γκρίνει εμείς. Όταν μιλάμε λοιπόν, και έχω μιλήσει με αγρότες, μίλησα και στο φόρουμ ε, για τη γεωργία και τα είπα έξω από τα δόντια, είπα ποιες είναι οι ανησυχίες μου και όταν εγώ μιλώ για γεωργία είπα δεν σημαίνει ότι όλη η γεωργία είναι επιζήμια. Υπάρχουν και καλές πρακτικές, υπάρχουν και κακές πρακτικές. Εγώ απλά θέλω να πω ότι δεν πρέπει να συνεχίσουμε να επιδοτούμε τις κακές πρακτικές. Αντίθετα, να αρχίσουμε να δίνουμε κίνητρα, να παρακινούμε ε, για τις ε, καλές πρακτικές. Καλύτερα προσπαθήσουμε να επιδοτήσουμε τις καλές πρακτικές αντί να επιδοτούμε τις επιζήμιες, τις κακές πρακτικές. Ναι, συνεργάζομαι σε πολύ καλό επίπεδο με τον Στάνφο Φερχόγγεν που κατανοεί το πρόβλημα και μάλιστα έχει χρηματίσει κατά το παρελθόν υπουργό περιβάλλοντος στη χώρα του, άρα γνωρίζει πολύ καλά και το περιβάλλον. Συμφωνούμε και οι δύο ότι θα πρέπει να συμμετέχουν οι αγρότες, ε, ο τομέας, ο γεωργικός κλάδο πρέπει να συμμετέχει. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα σχέδιο δράση που δεν θα προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα βασικά αιτία της ε, υποβάθμισης της βιοποικιλότητας. Ε, σε ό,τι αφορά την αρινή θύρα δεν είμαι υπέρ και νομίζω ότι φέτος για πρώτη φορά καταφέραμε να έχουμε απαγόρευση του κυνηγιού στην την Άνοιξη και στη δική μου χώρα που την ξέρω πολύ καλά αλλά ξέρετε απογοητεύτηκα όταν είδα κάτι ε, στην, ε, σε μια έκθεση για τα είδη τα οποία ε, τα κυνηγούν την, το φθινόπορο. Υπάρχει αυτή η πρόταση να σταματήσει το κυνήγι την άνοιξη, αλλά δεν συνεχίζεται και γίνεται και τον... το φθινόπωρο. Πώς θα γίνει για κάποια είδη. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία που λέτε ότι πήρε, ε, είχε πιο διάρκεια σε πιο πολύ από όσο έπρεπε. Ναι, πράγματι έγινε αυτό. Περιμέναμε και οι πολίτες να έχουν μια πολύ καλή ε, συμμετοχή. Για το νερό μιλάω. Ξέρετε ότι ήταν η μεγαλύτερη διαβούλευση από πολίτες. 500.000, δηλαδή μισό εκατομμύριο email πήραμε. Για να μην πω τι επιστολές πήραμε από τα κράτη-μέλη, από υπουργούς, ΜΚΟ, βουλευτές. Άρα φυσικά θέλουμε να το ε, φέρουμε σε πέρας. Αλλά εγώ προχωρώ πέραν της εντολής μου. Θα μπορούσα να μην ε, έχω προχωρήσει, γιατί δεν περιλαμβάνω ε, αυτό το χαρτοφυλάκι στο σχέδιο δράση, αλλά εγώ προχώρησα. σε ό,τι αφορά το γαλάζιο παράθυρο που κατέρευσε, είμαστε συγκλονισμένοι. Το είχαμε και λογότυπο στη διάσκεψή μας για τους ωκεανούς. Δυστυχώς αυτό είναι μια από τις περιπτώσεις που η φύση καταστρέφει τη φύση. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι να αποφευθεί η καταστροφή αυτή, αλλά είναι σίγουρα μεγάλη πολύ για το δάσος στην Πολωνία. Πράγματι, υπάρχει διαδικασία επί παραβάση. Πρόσφατα όμως με ενημέρωσε με επιστολή του ο ότι είχαν ένα τροποποιημένο διαχειριστικό σχέδιο με πρόθεση να ξεκινήσουν να αυξάνουν την υλοτόμηση και πήραμε πρωτοβουλίες. Εγώ έστειλα αμέσω επιστολή ζητώντας από τον Υπουργό να αναστείλει άμεσα τις δραστηριότητες υλοτομίας. και παρότι προσφερθήκαμε να συζητήσουμε την τροποποίηση του σχετικού νόμου, δεν έγινε δεκτή η προσφορά μας. αλλά θα προχωρήσουμε στην επόμενη φάση της διαδικασίας παραβάση. Για το νερό, Λίν, πρώτα απ' όλα να πω ότι η θέση της Κομισιόν είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη και την έχουμε εκφράσει επανειλημμένως και εγώ προσωπικά απαντώντα σε ερωτήσεις βουλευτών και στην Επιτροπή Προγραμμόνων και σε μία επιστολή στον κ. Σάιμον Κόβεν και πρόσφατα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή προφορικά. Δεν θέλω να μπω λοιπόν σε λεπτομέρειες. Θα πρέπει λοιπόν η Λαϊκή Κυβέρνηση να κάνει μια πρόταση που θα σέβεται την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, γιατί αυτός είναι ο στόχος, ο σεβασμός των αρχών ανάκτησης του κόστους. Για τις υπηρεσίες και την επιστολή αυτή, αυτά που αναφέρατε, Εγώ απάντησα στην επιστολή της κυρίας Μπόιλ ε, φέρε σε αυτή την επιστολή σε αυτή την εβδομάδα. Δεν έχω να πω τίποτε παραπάνω, πέραν του ότι εξετάζουμε το θέμα και υπάρχει σχετική έρευνα την οποία θα ε, μελετήσουμε. Εγώ έδωσα εντολή σε όλο μου το προσωπικό να υποστηρίξει την έρευνα της ε, Ευρωπαίας Δημοσιολαβήτριας για το θέμα αυτό. Κατά πόσον τώρα ήταν εύκολη όχι εντολή μου. Μου τρέψει να διαφωνήσω για την κοινωνική πολιτική. Ναι, τη μεταρρύθμιση αυτή θα την παρακολουθήσουμε εκ του Ο Επίτροπος Χόγκαν ε, είναι ο αρμόδιος Επίτροπος. Ήδη έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις μεταξύ των συναδέλφων μου και των συναδέλφων του γραφείου του κ. Χόγκαν και με άλλες υπηρεσίες επίσης. το σχόλιο του προκάτοχος με έκανε ότι μπορούσε για να είναι πράσινη η ΚΑΠ. Ναι, αυτό που λέμε σήμερα είναι ότι πράγματι το πρασίνισμα υποτίθεται πρέπει να γίνει με την ε, κοινή γεωργική πολιτική, δεν έγινε. Άρα πρέπει να συνεχίσω από πού άφησε τα πράγματα ο προκατοχό μου. Και να συνεχίσω να απευθύνω έκκληση να έχουμε πρασίνισμα της κοινή γεωργικής πολιτικής και ελπίζω να ληφθεί αυτό υπόψη. Και χρειαζόμαστε και τη δική σας υποστήριξη. Δεν μπορούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να μείνουν στο ίδιο στρατόπεδο. Είναι πολύ σοβαρή υπόθεση το Dieselgate. Είναι θέμα της ποιότητας της ατμόσφαιρας. Τα είπα αυτά και στις αρχές μου δηλώσεις. Αλλά φυσικά και η ατμοσφαιρική ρήπανση σκοτώνει μας προβληματίζει και είπαμε ότι θέλουμε να έχουμε τις μισές τέτοιες επιπτώσεις με το 2031 στόχος και έχουμε και το πρόγραμμα Cleaner για την Ευρώπη καλύπτει αυτούς τους στόχους και αυτό είναι και στην οδηγία NET που πέρσι εγκρίθηκε οπότε θα πρέπει όμως και αυτή να εφαρμογεί έχουμε και τις οδηγίες που άρχισαν να τρέχουν το 2015 που ονομάζονται LCP και ξεκινήσαμε μια σειρά επαφών με τα κράτη-μέλη για την ατμοσφαιρική ρήπανση και ξεκινήσαμε με την ε, Ιρλανδία για το πρόγραμμα Cleaner και ε, μετά θα ακολουθήσει Λουξεμβούργο και Ουγγαρία ούτως ώστε να υπάρξει περισσότερη συμμόρφωση αλλά και ανάληψη δράσης. Επίσης θέλουμε να υπάρξει και κύρωση του πρωτοκόλου του Γκότεμπεργκ ε, και γι' αυτό συνεργάζομαι με τη Μαλτέζικη Προεδρία. όσον αφορά τι ε, περιβαλλοντικέ επιθεωρήσει, και αυτό βρίσκεται στο θεματολόγιό μα, αλλά και η εύκολη πρόσβαση στην ε, δικαιοσύνη. Και αυτό μα απασχολεί. Θα το παρουσιάσουμε γι' αυτό. Επίσης, να σας προσθέσω θα το δώσω έξω κυρία Μαγκίνες ότι εξετάζουμε αυτά τα θέματα όσον αφορά το τι νομοθεσία, τι πτώση η νομοθεσία η κοινοτική για την ελληνική πολιτική. Είχαμε επί δυόμιση ώρα, δυόμιση ώρα συγγνώμη, συζήτηση ε, για τα θέματα αυτά στο Ιρλανδικό Κοινοβούλιο, ξέρετε. Είχα μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση, λέει η κυρία Μπόιλαν. Από τότε που αναγίνησε το θέμα εκείνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο έχουν πέρασει τόσα χρόνια. Ναι, πρόκειται για αυτή την πρωτοβουλία των πολιτών για την πρόσβαση στο νερό. Πάνω από ένα εκατομμύριο είχαν προσυπογράψει. Και εκεί γίνεται πρόοδος. Το, το εξετάζει ο αρμόδιος συνάδελφος. Well, thank you. Η πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε και τώρα οι υπόλοιποι συνάδελφοι που έχουν σειρά, η να Μποναφέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και κύριε Επίτροπε που σήμερα ήρθατε να μας μιλήσετε. Άκουσα από τους προλαλήσαντες το πόσο χρειάζεται να αρθεί αυτό το, χάσμα μεταξύ ε, γεωργίας και περιβάλλοντος. Δεν θέλω να είμαι αιρετική, αλλά νομίζω ότι το πρόβλημα, η πρόκληση που έχουμε και εμείς και εσείς είναι άλλο κενό, άλλο χάσμα μεταξύ περιβάλλοντος και βιομηχανίας. Το χάσμα που χωρίζει αυτούς τους δύο τομείς, οπότε ε, είπαμε ότι το περιβάλλον θα πρέπει να συνδυαστεί με την ε, άνοδο του ΑΕΠ, της απασχόλησης κλπ. Επομένως τέτοιου είδου συνέργεια χρειάζεται και βέβαια είναι πολύ σημαντική η κυκλική οικονομία στη σχετική μας ε, επιχειρηματολογία όχι μόνο για ανάκτηση πρώτων υλών που βρίσκονται σε σπάνιδα, αλλά και κοστίζουν και πολύ. Και αυτό θα γίνεται από τα απόβλητα, αλλά επίσης να μπορούμε να έχουμε πιο αποτελεσματικούς παραγωγικούς κύκλους και πιο βιώσιμους για κάποια προϊόντα λοιπόν τα οποία επιδέχονται τέτοια βιωσιμότητα. Όπως είπατε θα μιλήσουμε για την κυκλική οικονομία, για τις τέσσερις ε, οδηγίες στο Στρασβούργο, σε οδηγίε για τα απόβλητα. Θεωρώ, επίτροπε, ότι το να περάσουν οι εκθέσεις μας ε, για αυτές τι τέσσερι οδηγίε. δεν θα είναι το τέρμα της διαδρομή, αλλά η αφετηρία της για την πορεία προ την κυκλική οικονομία και επίσης θα πρέπει να βοηθηθούμε από τα όσα προβλέπει ήδη το πρόγραμμα δράσης. πρώτη δράση είναι η στρατηγική για τα πλαστικά υλικά, κάποια ευαίσθητα υλικά. Που όταν μιλούμε για την θαλάσσια ρήπανση, τα αναφέρουμε συχνά. Αλλά υπάρχει το θέμα βέβαια της ανακύκλωσής τους αυτών των υλικών. Αλλά θα πρέπει να εμπλακούν και οι σχετικές βιομηχανίες που παράγουν το πλαστικό και να εμπλακούν στην ε, προώθηση βιοπλαστικών. Πέραν των ανακοινώσεων επομένω, θα πρέπει να υπάρξουν και κανονικά νομοθετήματα σχετικά. Κάτι άλλο μα είπατε για την ανακύκλωση του, του, του νιδάτων που χρησιμοποιούνται στην γεωργία κλπ. Ξέρουμε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό και είπαμε ότι μέχρι τέλος χρονιά θα υπάρξει ένα νομοθέτημα, θα κάνετε κάτι, ίσω μάλλον τις διακοπέ, διακοπές. Εγώ φυσικά είμαι υπέρ όμως κυκλοφορούν κάποιες φήμες για το ότι αυτή η οδηγία δεν θα καλύψει πολλά κράτη-μέλη. Όμως, σχετικά με την αποτελεσματική χρήση των ε, πόρων θα είναι πάρα πολύ σημαντικό βήμα πρόοδου αυτή η οδηγία για την ε, πολλαπλή ας πούμε χρήση των υδάτων αυτών της γεωργίας. και είπαμε ότι χρειάζονται επενδύσεις αλλά πώς θα υποστηρίξουν αυτό μας το όραμα οι χώρες που θα ανήκουν στην δεύτερη ή τρίτη ταχύτητα στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ, η κυρία Σουίτσα. Ευχαριστώ. Έχω ένα συγκεκριμένο ερώτημα, μια και ασχολείστε και με το περιβάλλον, την προστασία της θάλασσας και της ε, ποιότητας του αέρα η Κροατία είναι χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τηρεί όλα τα κριτήρια και τις προδιαγραφές ε, για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά έχουμε πρόβλημα με την τήρηση αυτών των προδιαγραφών από, τους, ε, από τις γειτονικές χώρες που δεν σέβονται ακριβώς αυτές τις, ε, τα κριτήρια του, τα περιβαλλοντικά και γι' αυτό έχουμε πρόβλημα. Ένα δηληστήριο στην περιοχή Μπόσας και Μπρότ δημιουργεί τεράστια ατμοσφαιρική ρήπανση. Επίσης έχουμε απόβλητα που από την Αλβανία ε, χύνονται στην Αδριατική θάλασσα. Οπότε έχουμε μεγάλη ρήπανση της Αδριατικής θάλασσας που επηρεάζει κυρίως τις ακτές της Κροατίας. Ε, είχαμε τη, ε, τις συστάσεις από τη Σύμβαση της Βαρκελόνης και έχουμε και την οδηγία που εμποδίζει ε, τέτοια ρήπανση και επιβάλλει έλεγχο. Ε, πώς θα φροντίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε οι χώρες που προσβλέπουν σε προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένταξη θα τηρήσουν τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές εφόσον έχουν υπογράψει ή πρέπει να υπογράψουν τέτοιου είδους περιβαλλοντικές συμφωνίες. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ. ευχαριστώ και ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που ήρθατε. Δεν θα σας εκπλέξει φαντάζομαι που και εγώ έχω ερωτήσεις ε, για τους ωκεανούς όπως πάντα. Ευχαριστώ καταρχήν για την ανακοίνωσή σας για την διακυβέρνηση των ωκεανών. Πολύ σημαντική. Ζητήσατε παγκόσμιους, ε, παγκόσμια προγράμματα για την ε, διακυβέρνηση των ωκεανών και των θαλασσών και ελπίζω στον το 2020 να ληφθούν υπόψη οι ερευνητικές προσπάθειες για τις θάλασσες και τους ωκεανούς και να είναι μονίμως ε, σημαντική προτεραιότητα. Ε, παρόλο που είναι ρητορική ερώτηση, δεν πιστεύετε ότι θα πρέπει να διευρύνουμε τις ε, αρμοδιότητες Επιτροπής Αλληλείας ώστε να είναι αρμόδια για οτιδήποτε αφορά τις θάλασσες και τους ωκεανούς. Να γίνει όχι Επιτροπή Αλληλείας μόνο, αλλά και Επιτροπή Αλληλείας και Θάλασσας. Επίσης, η γενική σας διάθεση δηλαδή ε, για την αλληλεία να περιλαμβάνει και τη θάλασσα. Επειδή το, οι ωκεανοί είναι θέμα οριζόντιο, θα πρέπει να υπάρχει μια ομάδα που να συντονίζει τις εργασίες των ε, γενικών διευθύνσεων που εφαρμόζουν πολιτικές που επηρεάζουν τους ωκεανούς. Επίσης, ε, μιλήσαμε για τα πλαστικά, αλλά τα μικροπλαστικά είναι επίσης πρόβλημα. Ε, τέτοια κατάλοιπα τα έχουμε βρει στο αλάτι που προέρχεται από τις αλικές, σε ψάρια, σε φυτά. Πώς θα καταπολεμήσουμε λοιπόν ε, τέτοια μικροπλαστικές ε, ουσίες που προέρχονται από υποδήματα, ρούχα, ε, ελαστικά. Πώ θα μειώσουμε λοιπόν την παραγωγή των μικροπλαστικών καταρχήν. Ευχαριστώ κύριο Σέκ. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο που είναι εδώ σήμερα στον Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γερμανία, στην Ολλανδία και στη Γαλλία, αλλά και στις ακτές της Νέας Ζηλανδίας με βάση τα μέσα ενημέρωσης υπάρχουν εξοκύλοι φάλαινες και οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν το λόγο γιατί έχουν φύγει από τις συνήθεις ε, ε, περιοχές ε, οι φάλαινες αυτές μάλλον λόγω των πλαστικών και των δικτυών που βρίσκονται στα νερά. Βλέπουμε λοιπόν ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ρήπανσης των ωκεανών από το πλαστικό ε, και χαίρομαι που αναλαμβάνει σχετική ε, πρωτοβουλία η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε όμως και τα σόναρ που δημιουργούν η χορύπανση στους ωκεανούς και έχω μια ερώτηση κατά πόσον ε, η Κομισιόν έχει σχέδια, γιατί βλέπουμε πολύ αρνητικά φαινόμενα, αν, αν υπάρχει δυνατότητα να γίνει μια γενική ε, έρευνα σε ό,τι αφορά την ε, ηχορύπανση και σε ό,τι αφορά τη βιοπικιλότητα είναι τελευταίο ερώτημα. Θεωρείτε, είπατε και τη θαλάσσια βιοπικιλότητα πάρα πολύ σημαντική. Υπάρχει αύξηση του πληθυσμού, αλλά και πάλι τα πράγματα μπορούσαν να ε, γίνουν αρνητικά στο μέλλον. Έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμη. Ε, ξέρουμε ότι υπάρχει κοινή φαλενών ε, στην Ιαπωνία. Υπάρχει σφαγή των βαλενών. Τι, φαλενών. Τι μέτρα θα πάρετε. Ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Uh, no, Madam Ευχαριστώ κυρία Όκεν. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και τον Επίτροπο που ήρθε. Νομίζω ότι θα πρέπει να γιορτάσουμε γιατί είχαμε ένα θετικό μέτρο. Ε, υποσχεθήκατε εδώ ότι θα συνεχίσετε διαδικασία επιπαραβάσεις βάρος της Πολωνίας για την συνέχιση της υλοτομίας στο δάσος που αναφέρατε. Επιτέλους, έχουμε κάτι απτό να γιορτάσουμε και να αναδείξουμε, όχι απλώς ε, υποσχέσεις, στάματα και ωραία λόγια. Συνεχίζοντας αυτά που είπε η Σιμώνα Μποναφέ για τη στρατηγική μας για τα πλαστικά. Δεν αρκούν οι ανακοινώσεις. Θέλουμε νομικά δεσμευτικές πράξεις. Ε, το ζητούμε εδώ και πολύ καιρό. Συμφωνώ λοιπόν, θα πρέπει να είμαστε πιο δραστικοί απέναντι στα πλαστικά. Και τέλος, τι γίνεται με τη νομική σας υποχρέωση να υποβάλλετε μια πρόταση για τον περιορισμό των πλαστικών σακουλών. είπατε, θα πρέπει να έχουμε μεθόδους υπολογισμού αυτών των πλαστικών ε, σακουλών. Και ήσασταν σαφή στη συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υποσχεθήκατε ότι θα αναλάβετε το καθήκον αυτό και θα τηρήσετε αυτή την νομική υποχρέωση. Ε, την περιμένουμε επιτέλους αυτή την πρόταση. Και ένα άλλο συναφές πρόβλημα που περιλαμβάνεται στη σχετική οδηγία. Τα βιοαπικοδομήσιμα και μάλιστα έχουμε σχετικές ε, εκστρατείες στην Ισπανία, στην Αφρική, στην ε, ε, Κύπρο. Ακόμη και στη Δανία έχει φτάσει αυτή η εκστρατεία. Θα πρέπει να γίνει μια έρευνα για τις για την ανάγκη να επιβληθεί επιτέλους απαγόρευση γιατί μιλήσατε για την α, παρουσία πλαστικών στη γεωργία. Αλλά τι γίνεται με την παρουσία των μικροπλαστικών παντού. Οπότε θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να εφαρμοστεί η σχετική πρόταση. Ελπίζω να απαντήσετε ξεκάθαρα. Γιατί ακόμη και τα βιοδομήσιμα υλικά έχουν επιβλαβεί ουσίε. Ελπίζω να με προσχεθείτε ότι σε λίγε μέρε, ο Σονόπου θα τη σχετική πρόταση. Ο κύριο Φαρία. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που ήρθατε. Θα μίλα για την ε, διακυβέρνηση της υπόθεσης των ε, ωκεανών με και εισηγητή σχετικού κειμένου αλλά ήδη φύγει το ζήτημα και με καλύψατε μετά όσο είπατε και σας ευχαριστώ και γι' αυτό. Τώρα κάτι άλλο όμως, κάτι άλλο. Να σας τα πω στα πορτογαλικά. Κύριε Επίτροπε, ε, πολύ κοντά στα πορτογαλικά σύνορα δημιουργείται ε, μία αποθήκη πυρηνικών αποβλήτων σε ισπανικό έδαφος, αλλά πολύ κοντά στα πορτογαλικά σύνορα. Χωρίς μάλιστα να έχει προηγηθεί διαβούλευση με τις πορτογαλικές αρχές. Και έχουμε και άλλα τέτοια προγράμματα και σχέδια. Για να μην μιλήσουμε για την ε, πρόθεση της ισπανικής κυβέρνησης να ξανανοίξει στο Μπούργος ένα παλιό πυρηνικό εργοστάσιο πολύ κοντά λοιπόν ε, ε, στην, ε, στον ποταμό Ντόουρο. Και έχουμε και άλλα τέτοια ισπανικά σχέδια, πολύ κοντά στην Πορτογαλία, που είναι επιβλαβή για το περιβάλλον, όπως είναι η εξόριξη ουρανίου, που θα ξεκινήσει στη Σαλαμάνκα, ή ένας σταθμός επεξεργασίας ουρανίου στο Ρετορδίλιο. Όλα αυτά λοιπόν τα επιβλαβή για το περιβάλλον προγράμματα α, της Ισπανικής κυβέρνησης δεν είχαν καν κοινοποιηθεί στην Πορτογαλική αρχή. Δεν θεωρείτε ότι παραβιάζουν την οδηγία 2000 κάθετο 42 του Ιουνίου του 2000 που σε τέτοιου είδους προγράμματα που έχουν διασυνοριακές περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα πρέπει να κοινοποιούνται στην ενδιαφερόμενη κυβέρνηση. Στις 11 Μαρτίου, το επόμενο Σάββατο λοιπόν, θα έχουμε την θλιβερή επέτειο της ε, πυρηνικής καταστροφής της Φουκουσίμα. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει τα μέτρα τους τα, κράτη-μέλη να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους και θα θέλαμε ε, ε, να ξεκινήσουν τέτοιες ε, διαδικασίες επί παραβάση σε περίπτωση που τα κράτη-μέλη δεν πληρούν τις υποχρεώσεις τους. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν τα επιβλαβή περιβαλλοντικά προγράμματα της Ισπανίας που παραβιάζουν και την οδηγία την, της 42 του 2001 και την ανάγκη προηγούμενης εκπόνησης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ελπίζω λοιπόν να, να λάβετε υπόψη όλα αυτά τα, όλες αυτές τις παραβιάσεις και να λάβετε μέτρα. Μπορείτε και με άλλους εσωτερικούς διάβλους να υποβάλλετε προ, Ερωτήσει προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν χρειάζεται να εξαντλείτε τώρα όλο σα τον χρόνο. Ο Πρώτα, πρώτα, μας ε, αναφέρεται σε σχέση με την έκθεση της κυρίας ε, Μποναφέτη θα γίνει με την ε, οδηγία για την κυκλική οικονομία και έχετε δίκιο σε αυτό που μας είπατε ότι πρόκειται για πολύ σημαντικό διακύβευμα πρόκειται για στροφή Πρόκειται για αλλαγή του οικονομικού προτύπου. Υπάρχει το θέμα βέβαια της διασπάθησης των τροφίμων. Ε, αυτό μας το θίξατε παρά το ότι υπάρχει στην, ε, κάποια τροπολογία που ψηφίζει στην Επιτροπή μας. 89 τόνοι διασπαθήσεων κάθε χρόνο. Και αν μπορούσαμε να φτάσουμε τα 120 εκατομμύρια τόνους του 2020 είναι τρομερά αυτά τα νούμερα και χρειάζεται επομένω ευρωπαϊκό στόχο. Και το ότι δεν ε, έχει τεθεί αυτό ο στόχο είναι ανεύθυνη πολιτική. Γι' αυτό και σα ερωτώ, εάν σε σχέση με αυτή την τροπολογία που εγκρίθηκε στην Επιτροπή μα, θέλετε μέσω του τριλόγου να δεχθείτε αυτή την τροπολογία. Κάτι που ακόμα δεν έχει γίνει. Ε, όπως μας ε, τονίσατε, θα ζητήσετε από πέντε χώρε να μπουν σε αυτό το πρόγραμμα για να μειώσουν τι εκπομπέ του διοξιδίου του αζότου και μετά από ορισμένου μήνες είχαμε επιστροφή αυτών των μεγάλων χωρών. Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία. Οπότε βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ η ρήπανση από αυτές τις χώρες του τελευταίους μήνες. Άρα το πράγμα επήγε. Μήπως θα πρέπει να υπάρχει κάποιο είδους ε, δεσμευτική πολιτική και να επιβάλλονται και κυρώσεις προς αυτές τις χώρες. Κυρία Γκούτελαντ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ξέρω ότι πιέζει ο χρόνος ε, και δεν θα ρωτήσω κάτι που ήθελα να ρωτήσω γιατί το έθεσε πάρα πολύ ολοκληρωμένα η Σιμώνα Μποναφή για την κυκλική οικονομία. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να φυγεί. Ε, ε, με την ευρύτερη διάσταση ε, στο έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά εντάχει να σας πω κάτι για τις μέλισσες, οι οποίες στην Ευρώπη πεθαίνουν. Και όχι μόνο στην Ευρώπη. Σας το έχω ήδη προαναφέρει. Θα ήθελα να μου πείτε εσείς στην Επιτροπή πώς θα το αντιμετωπίσετε το πρόβλημα. Γιατί υπάρχουν πολλές αιτίες που δημιουργούν αυτό το φαινόμενο ένα εκ των οποίων είναι και τα ζυζανιοκτώνα. Θα πρέπει να σώσουμε τις μέλισσες. Για πέστε μας τι πρεσβεύετε. Τώρα κάτι άλλο για το φινικέλαιο και για τη στροφή προς μια βιώσιμη παραγωγή. Πώς θα εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχει αποψήλωση των δασών στις χώρες παραγωγούς. Όπως γνωρίζουμε χρησιμοποιείται για τα είδη διατροφής αυτό το έλαιο, αλλά και στα βιοκαύσιμα το φινικέλαιο. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εξασφαλίσει ότι δεν θα πρέπει τα δύο να περιέχουν στοιχεία μη βιώσιμα όπως το ε, φινικέλο να είναι κάτι πιο φιλικό στο περιβάλλον και στο κλίμα αυτό που χρησιμοποιείται δηλαδή το φινικέλο να μην παράγεται με μη βιώσιμο τρόπο και μετά να χρησιμοποιείται στα τρόφιμα και στα βιοκαύσιμα. καύσιμα. Ε, Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε και τώρα έχει το λόγο η κυρία Γκαρθία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πιέζει ο χρόνο οπότε... Κι εγώ, κι εγώ, λέει ο κύριο Ζωρίνιο, κι εγώ έχω ζητήσει το λόγο. Α, έχετε μήπω σε σειρά. Πάλι, η κυρία Γκαρθία. Είπα ότι πιέζει ο χρόνος και θα ήθελα να σας ρωτήσω Δύο, δύο ερωτήσεις έχω συγκεκριμένα σε επίτροπε. Πρώτα πρώτα, σε σχέση με αυτό το στόχο που είπατε και ότι πώς σας ενδιαφέρει για την μείωση χρήση του καδμίου συγκεκριμένα. Σας ρωτάω, θεωρείτε ότι σε αυτή την πρόταση της Επιτροπής ε, σύμφωνοι για το στόχο σας ε, γίνεται μέσα στα πλαίσια που έχει θέσει και ορίσει η πρότασή σας να συνεχίσουν οι εισαγωγές φωσφορούχων βράχων από το Μαρόκο, πετρωμάτων τέλο πάντων. Και επίσης για πέστε μας, γίνεται να σταμα... γιατί είναι πολύ σημαντικές αυτές οι εισαγωγές. Τώρα όσον αφορά τα λοιπάσματα στην άγκρη, είπαμε ότι θα πρέπει να δούμε πώς θα βελτιώσουμε τα οργανικά ή βιολογικά προϊόντα. Εσείς πώς νομίζετε ότι θα πρέπει για τα αζωτούχα να εφαρμοστεί η οδηγία και να έχουμε καλύτερη παραγωγή βιολογικών προϊόντων χωρίς να έχουμε λιπάσματα χημικά γίνεται αυτό στα πλαίσια της οδηγίας για τα αζωτούχα. Τα συζητήσαμε, είπαμε, στην Επιτροπή Γεωργίας, τα σχετικά με τα λοιπάσματα. Ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ζωρίνια. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Έχω μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση. Το σχέδιο για την πυρηνική ενέργεια του 2016 προβλέπει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε 88 παροπλισμένα πυρηνικά εργοστάσια που δεν έχουν όμως ε, κλείσει. Είναι απλώς ανενεργά και τα περισσότερα πυρηνικά εργοστάσια στην Ευρώπη έχουν ξεπεράσει την κανονική διάρκεια ζωή τους. Αυτό δημιουργεί τεράστιες προκλήσεις. Και μάλιστα έχουμε 100 χιλιόμετρα από τα, ευρωπαϊκά, από τα σύνορα κοντά στο Τάγο στην Ισπανία που διακυβεύουν την ασφάλεια. Πότε σκοπεύουν οι Ισπανοί επιτέλους να παροπλήσουν και να κλείσουν το εργοστάσιο. Θέλουμε ένα ευρωπαϊκό σχέδιο εκτάκτου, το ανάγκης για να αντιμετωπίσουμε τα πυρηνικά εργοστάσια που είτε πρέπει να κλείσουν είτε βρίσκονται στο τέλος της ζωής τους ε, και θα πρέπει να παροπλιστούν. Ευχαριστώ. Τελευταίος αλλά εξίσου σημαντικός ο κύριος Καπούτο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εσάς κύριε Επίτροπε που ήρθατε και που είσαστε πάντοτε πρόθυμος να μας μιλήσετε. Βεβαίω και δεν και να επαναλάβω τις ερωτήσεις που έχουν προηγηθεί από τους συναδέλφους. Πάρα πολύ καλά τα είπε για την κυκλική οικονομία η Σιμώνα Μποναφέ. Την ενδιαφέρει το θέμα. Τώρα, όμως θέλω να σταθώ στο θέμα το οποίο εσείς αναφέρατε, αλλά πάρα πολύ λίγο. Δηλαδή όσον αφορά την ατμοσφαιρική ρήπανση ε, τις ιστορικές και εξωτερικές. Είναι πολύ σημαντικό κίνδυνος αυτός και για το περιβάλλον και για την ανθρώπινη υγεία, γιατί έχουμε κάποιες μελέτες της Ευρωπαϊκής Υγείας και λένε ότι έχουμε θανάτους 6 εκατομμυρίων ανθρώπων εξ αυτού του λόγου και κυρίως κάποια βρέφη τα οποία παραβλάπονται. Και αυτή η έκθεση του Οργανισμού Υγείας. Θα μπορούσε να είναι χρήσιμη πηγή πληροφοριών, θα μπορούσε να είναι μια αφετηρία για τις ευρωπαϊκές πολιτικές και για τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τα νομοθετήματα τέλος πάντων. Το έχει λάβει αυτό υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει λάβει υπόψη την έκθεση αυτή και δύναμη αυτού του υλικού θα προχωρήσετε σε αναθεώρηση των ισχυών των κανονισμών Πήγαινε γενικότερα της νομοθεσίας σχετικής με το θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Καμπεθόν Ρουίθ. Ένα σχόλιο και μια ερώτηση. Μάλλον δύο ερωτήσεις. Καταρχάς το σχόλιο για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης που ανακοινώσετε για την εφαρμογή της οδηγίας για τα ενδιατήματα και την Α λέτε ότι καλύτερο είναι να μην έχουμε μια οδηγία αλλά να εφαρμόσουμε την υφιστάμενη καλύτερα. Έχουμε κάποια καθυστέρηση. Ελπίζω το σχέδιο δράσης να βοηθήσει ε, στην εφαρμογή της οδηγίας. Αλλά να μην γίνει φραγμός, να μην γίνει ένα γραφειοκρατικό εμπόδιο και σίγουρα να μην μειωθούν οι στόχοι της οδηγίας. Το σχόλιο μου δηλαδή ουσιαστικά είναι ότι το σχέδιο δράσης με τους στόχους του έχει ε, ως σκοπό να βοηθήσει την ε, υλοποίηση των στόχων και να μην γίνει ε, αιτία να έχουμε μικρότερη ακόμη εφαρμογή υλοποίηση. Είπατε, ρωτήσατε αν εμείς θα καταθέσουμε ψήφισμα. Δεν ξέρω αν χρειάζεται κάποιο μήνυμα ή αν μπορούμε να σας στηρίξουμε ε, να ακολουθήσουμε μια συγκεκριμένη γραμμή στο Κοινοβούλιο. Και για την ε, ερώτηση για το νερό. Ο κύριος Γιούνκερ, πρόεδρος της Κομισιόν, έχει μιλήσει για την νομοθετική οικονομία Δηλαδή να μην γίνεται πολύ νομοθετική δραστηριότητα. Όμω το νερό θα μπορούσε να είναι ένα από του ε, τομεί, μία από τι πρωτοβουλίες που χρειάζεται να αναλυφθούν. Στηρίζουμε λοιπόν ε, την πρόταση γιατί έχει υπάρξει μεγάλη λαϊκή κινητοποίηση για το θέμα αυτό. Είπατε ότι τα σκέφτεστε, αλλά τι συγκεκριμένα σκέφτεστε. Σκέφτεστε ένα είδος νομοθετικής πρωτοβουλίας για αυτό το τόσο σπάνιο αγαθό που πρέπει να το διαφυλάξουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Είδατε τι ζωηρό ενδιαφέρον να προκαλέσατε με την παρουσίασή σας. Ε, η πλειάδα ερωτήσεων, θετικό το κρίνω. Φυσικά θα προλάβετε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις διεξοδικά. Αλλά θα βρούμε κάποιο τρόπο είτε σε άλλη ανταλλαγή απόψεων, είτε γραπτός για να δώσουμε απαντήσεις. Εσείς τώρα επικεντρωθείτε στα πιο ουσιώδη κατά τη γνώμη σας. Θα βάλω τα δυνατά μου για να απαντήσω στις περισσότερες ερωτήσεις. Αν δεν προλάβω, θα σας στείλω τις απαντήσεις γραπτός. Σε ό,τι αφορά την, τις παρατηρήσεις κυρίας Μποναφέ, συμφωνώ ότι θα πρέπει να δούμε το χάσμα που υπάρχει μεταξύ βιομηχανία και περιβάλλοντος. Και η κυκλική οικονομία είναι εξαιρετικό παράδειγμα ότι με μία λύση μπορούμε να λύσουμε και περιβαλλοντικά και οικονομικά προβλήματα. Σε ό,τι αφορά το περιβάλλον και την οικονομία, έχουμε ήδη περίτρανες αποδείξεις ότι ο πράσινος κλάδος, ο φιλοπεριβαλλοντικός, ε, είναι πολύ στιβαρός και μάλιστα Κατά την κρίση ήταν από τους πιο θεκτικούς κλάδους οικονομίας ο πράσινος ε, τομέας και συνέχισε να μεγεθύνεται οικονομικά και να δημιουργεί θέσει απασχόληση ενώ οι άλλοι τομείς είχαν πάρει τον κατήφορο με την κρίση. Και φυσικά περιμένουμε με ανυπομονησία την ολομέλεια της επόμενης εβδομάδας στο Στρασβούργο και θα είμαι και εγώ παρόν εκεί. Η στρατηγική για τα πλαστικά την λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη, όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Και μάλιστα ε, παρέστηκε και ε, σε μία από τις περιβαλλοντικές συνεδριάσεις του G7 και ε, επιμείναμε να συζητηθεί αυτό στις συζητήσεις. Το θέμα των πλαστικών σε συνδυασμό με τα απορρίμματα στη θάλασσα και αυτό εξετάζεται και στις δικές μας γενικές διευθύνσεις. Η κυκλική οικονομία αφορά και τα χημικά, τι είδου χημικά χρησιμοποιούμε, σε τι δοσολογίες και η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία Πλαστικών μας υποστήριξε μέχρι στιγμής πολύ και θα συνεχίσει να το κάνει. Σε ό,τι αφορά την επαναχρησιμοποίηση των λιμάτων ε, του Είναι πολύ σημαντικό θέμα γιατί αυτό το νόημα έχει η κυκλική οικονομία. Να γίνεται αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων και η επαναχρησιμοποίηση του νερού που είναι από τα σημαντικότερα αγαθά του πλανήτη είναι βασικό στοιχείο της κυκλικής οικονομίας. Αλλά γενικώ η ανακύκλωση είναι σημαντικό τμήμα αυτής της κυκλικής οικονομίας και θα το αντιμετωπίσουμε αυτό σε επιμέρου πρωτοβουλίε. Η Σιμών αναφέρθηκε σε ορισμένε πρωτοβουλίε, πάντω στο πρόγραμμα εργασιών τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2010-2017 είχαμε τουλάχιστον πέντε αξιέπαινε πρωτοβουλίε που, περιλάβαμε και η στρατηγική για τα πλαστικά είναι μία από αυτές. Ε, καλύπτει και το θέμα της ανακύκλωσης και της, τα ποσοστά επαναχρησιμοποίησης των πλαστικών, επίσης διαρροή των πλαστικών στα τρόφιμα, στη θάλασσα και η θέλουμε να περιορίσουμε ε, την ε, απόλυτη εξάρτηση από τα πλαστικά κάποιων καυσίμων. Επίσης, είπαμε, θα ε, προσπαθούμε να εντοπίζουμε τέτοιες επικίνδυνες ουσίες, θα κάνουμε την επικαιροποίηση για την ανακύκλωση και προ... προτείνουμε απαλλαγή από τα από τις τοξικές ουσίες. Και μάλιστα θα έχουμε και ένα πλαίσιο για να καταμετρούμε την πρόοδο στην κυκλική οικονομία. Και μάλιστα θα έχουμε και νομοθετική πρόταση για τα ελάχιστα ποσοστά ε, για την επανεχρησιμοποίηση του, του ύδατος και θα ε, αναθεωρήσουμε και την οδηγία για το πόσιμο είδωρ. Και φυσικά με βάση την πρωτοβουλία των πολιτών ε, που είχε το, το ίδιο αντικείμενο. Η Σιμών επίσης μας ρώτησε τι επενδύσεις θα κάνουμε. Και μάλιστα ένα μεγάλο τμήμα των ταμείων του στρατηγικών επενδύσεων αφορούσαν την πράσινη οικονομία και δι' την κυκλική οικονομία. Αλλά έχουμε και τα κονδύλια του ορίζοντα 2020, 650, ευρώ, 650 ε, εκατομμύρια ευρώ. Καθόλου από ποσό που θα χρηματοδοτήσει την κυκλική οικονομία στα βιομηχανικά προγράμματα και σχέδια. Επίσης, ε, σε συνεργασία με την ΕΤΕΠ και άλλες τράπεζες, δημιουργούμε μια πράσινη πλατφόρμα για να διευκολύνουμε και να ενθαρρύνουμε, να παρατρύνουμε τη βιομηχανία να πραγματοποιήσει πράσινες φιλοπεριβαλλοντικές ε, επενδύσεις ή να επενδύσει στην κυκλική οικονομία. Σε ό,τι αφορά το θέμα της Κροατίας, έχουμε αρκετές δυσκολίες, αλλά έφυγε η κυρία που έθεσε την ερώτηση. Έχουμε διασυνοριακά προβλήματα και ζητήματα εκεί. Μερικά, μάλιστα, διασυνοριακά θέματα εμπλέκουν δύο ή τρία κράτη-μέλη ή εμπλέκουν κράτη-μέλη και τρίτες χώρες, γειτονικές πάντως χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και άρα εμπίπτουν στη στρατηγική γειτονία. Πάντως, όποιος και να εμπλέκουν αυτά τα διασυνοριακά θέματα θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τα διευθετήσουμε. Και αυτό κάνουμε. Και μάλιστα ο Επίτροπος Ιωάννης Αντεχάν, ο αρμόδιος για τη διεύρυνση, εμπλέκεται και αυτό στις συζητήσεις. Μιλήσαμε και για, και για τη μελλοντική συγχώνευση των Γενικών Διευθύνσεων Αλίας και Θαλασσών. Όταν ανέλαβε τη Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ των θαλασσών, ασχολούνται κατά 80% με την αλία και 20% με, τη, με τα θαλάσσια ζητήματα. Και είπα ότι θα πρέπει να ανατραπεί το ποσοστό, 80% να αφορά τη θάλασσα και 20% την αλία. δεν θέλουμε να περιορίσουμε το ενδιαφέρον της DG Mare για την αλία, αλλά να αναβαθμίσουμε το ενδιαφέρον της DG για τη θάλασσα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ομάδα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μια οριζόντια ομάδα για τους ωκεανούς, ο, οι ωκεανοί είναι οριζόντιο θέμα. Εμπίπτουν στα ε, χαρτοφυλάκια πολλών επιτρόπων. Ε, έχουν ε, επιπτώσει στο περιβάλλον, στις κλιματικές αλλαγές, ε, στη βιοπικιλότητα, στα τρόφιμα, γιατί είπαμε να σητήσουμε τον πλανήτη. Ο πλανήτης δεν σητίζεται μόνο από τη γεωργία, από το έδαφος, αλλά και από τους ωκεανούς. Γι' αυτό είπαμε ότι θέλουμε να συνεργαστούμε ε, και στην πρωτοβουλία μας για, την, ε, για τους ωκεανούς και να το έχουμε ως οριζόντιο ζήτημα πολλών πολιτικών. Γι' αυτό και με την ε, είπατε εκπρόσωπο συμφωνήσαμε να λάβουμε υπόψη τις τεράστιες εξωτερικές επιπτώσεις της διακυβέρνησης των ωκεανών και της Αρκτικής. Σε ό,τι αφορά τα μικροπλαστικά, είναι πολύ σημαντικό θέμα και κάποιες χώρες μέλη ήδη έχουν αναλάβει μονομερός δράση για τον περιορισμό της χρήσης τους. Εμείς ε, προς το παρόν προχωρούμε σχετικά επιφυλακτικά. Ήδη έχουμε αναθέσει την εκπόνηση μελετών για να ε, διαμορφώσουμε μια πιο εμπεριστατωμένη γνώμη και κατά πάσα πιθανότητα θα το συλλάβουμε υπόψη στη μελλοντική μας στρατηγική για τα πλαστικά. Εκεί που μιλούμε για microbees και άλλα θέματα, ε, υπάρχουν και άλλα κρίσιμα σημεία, όπως η σκόνη, ο κονιορτός που αφήνουν τα ελαστικά των αυτοκινήτων στους δρόμους μας. Αυτά τα σωματίδια από το κονιορτό είναι επίσης πολύ επικίνδυνα. Φαλαινοθυρία και βιοπικιλότητα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Ε, πολλές ε, ε, φάλαινες έχουν εξοκύλει και δεν γνωρίζουμε τα αίτια που τις έχουν οδηγήσει σε κάτι τέτοιο. Ίσως λόγω του περιορισμού της βιοπικιλότητας των ωκεανών. Για μερικά θέματα που συμβαίνουν στην ξηρά, εύκολα εντοπίζουμε τα αίτια, αλλά για φαινόμενα των ωκεανών, δυστυχώς δεν βρίσκουμε πάντα τα αίτια. Ακόμη και σε περίπτωση αεροπορικού ατυχήματο, ε, όταν συντρίβεται στην ξηρά, στο έδαφο, πολύ γρήγορα βρίσκουμε τα συντρίμια του. Αν όμω πέσει στη θάλασσα, οι έρευνε κρατούν πολύ περισσότερο και μερικέ φορέ χρειαζόμαστε τύχη για να το εντοπίσουμε. Το ίδιο ισχύει και με τα αίτια της, του φαινομένου αυτού που φέρνει όλο και περισσότερε φάρελε να εξοκέλουν στις ακτέ. Μπορεί να οφείλεται αυτό στην ηχορύπανση, στην ε, θαλάσσια ρήπανση. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να διαρευνούμε τα αίτια αυτού του φαινομένου. Και σε ό,τι αφορά τη φαλαινοθυρία εκ μέρους των Ιαπώνων, αυτό πάντα το τονίζω όταν πηγαίνω στην Ιαπωνία και διατρανώνω τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της φαλαινοθυρίας. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο δάσος στην Πολωνία, το ανέφερε και η κυρία Όγκεν αυτό που δεν εξήγησα προηγουμένως είναι ότι στείλαμε μέχρι και αντιπροσωπεία της Γενικής μας Διεύθυνσης ε, για να ε, διερευνήσει την κατάσταση και να δει τι συμβαίνει στο δάσος αυτό. Και μάλιστα και η UNESCO είχε στείλει αντιπροσωπεία. Και μάλιστα καταλήξαμε στα ίδια συμπεράσματα με την αντιπροσωπεία της UNESCO. Σε ό,τι αφορά τις πλαστικές σακούλες, νομίζω ότι το κάλυψα. Ήδη υπάρχει οδηγία για το θέμα αυτό και νομίζω ότι βρισκόμαστε στην ίδια γραμμή πλεύσης. Πρόκειται για οδηγία του 2015 και ήδη λειτουργεί, ήδη κάποιες χώρες την έχουν εντάξει του να τάξη και εφαρμόζεται. Πάντως παρακολουθούμε τα θέματα. Μίλησαμε επίσης και αυτές τις διασυνοριακές διαφορές και προστριβές που υπάρχουν και νομίζω ότι ο πρόεδρος Γιούνκερ έχει βοηθήσει να υπάρξει κάποια συμφιλίωση στην Ισπανία. Ελπίζουμε να βρεθεί τελικά κάποια λύση, αλλά συμφωνώ μαζί σας ότι όλοι θα πρέπει να συμμορφωθούν με την συμφωνία. Τρόσον αφορά τα πυρηνικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί, έχει υποσχεθεί να υπάρξει αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης και της ε, Ευρατόμ. Και εγώ, αλλά και ο συνάδελφος Κανιέται. Όσον αφορά τη διασπάθηση των τροφίμων και τα σχετική, σχετική ρήπανση και αυτό καλύπτεται από το όραμα της κυκλικής οικονομίας είναι παράλογο ότι έχουμε τόση διασπάθηση στην Ευρώπη. 40% αυτά το ποσοστό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πει στα κράτη-μέλη ότι θα πρέπει να εκπονήσουν ένα σχέδιο, ένα πρόγραμμα για το πώς θα διαχειριστούν την μείωση που θέλουμε, το στόχο που έχουμε τάξει για τη διασπάθηση των τροφίμων, ακριβώς όπως το θέλει και ο ΟΗΕ. Θα πρέπει όμως τα κράτη-μέλη σε τακτά διαστήματα να υποβάλουν κάποια έκθεση πρόοδο σε αυτό το μέτωπο για τις μέλισσες. Σας ανέφερα ότι αυτό καλύπτεται από το πρόγραμμα δράσης του ΡΙΦΙΤ για βιότοπους και πτηνά. Και όταν λέμε για επικονιαστές δεν είναι μόνο οι μέλισσες, είναι χιλιάδες ειδών. Πεταλούδες, πουλιά, μέλισσες και αυτό το ερευνούμε την ευρούμε το πώς με κάποιες μελέτες θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης το οποίο να καλύπτει ε, και τις μέλησες και όλους τους επικονιαστές. Οι μέλησες βέβαια είναι στο επίκεντρο προσπάθειας τώρα για το φινικέλαιο και στην αποψήλωση των ε, δασών και στην ε, επιδείνωση των δασών και της γης. Είναι ακόμη προτεραιότητά μα και έχουμε αναπτύξει δράση και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όχι μόνο, γιατί θα πρέπει να συνεργαστούμε με τις χώρες παραγωγούς. Προσωπικά πήγα στο Βιετνάμ, στην Ινδονησία και στη Μαλαισία, είχα επαφές εκεί και έχουμε θετική εμπειρία από το πρόγραμμα δράσης και από το σχετικό κανονισμό για την υλοτομία. Προσπαθούμε και προσπαθεί σκληρά η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα δάση. Στα πλαίσια των στόχων των αναπτυξιακών. Ε, βέβαια και η υποψήλωση των ε, δασών οφείλεται σε πολλές αιτίε, υπάρχουν διαφορετικές δυναμικές σε κάθε χώρα, άρα δεν μπορούμε να βρούμε ενιαία λύση για παντού. Και απαιτεί το θέμα συλλογική ανάληψη δράσης σε διεθνές και τοπικό επίπεδο. Όλοι εμπλακόμενοι να βοηθήσουν. Το 2016 η Επιτροπή έκανε κάποια μελέτη για το πώς θα ενταθεί η προσπάθεια να φρενάρουμε την αποψήλωση των δασών και αυτή η μελέτη θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2017. Και θα δούμε μετά τη μελέτη αν χρειάζεται ξεχωριστό πρόγραμμα δράσης. Και βέβαια αποτελεί πρόβλημα το φινικέλαιο διότι είναι ένα προϊόν που έχει πάρα πολύ μεγάλη απόδοση ανά εκτάριο και πολύ σημαντικό επομένω για τις χώρες ε, παραγωγούς. Όπως και στη Γεωργία γενικότερα έχουμε καλές και κακές πρακτικές. Δεν μπορούμε να τους βάλουμε όλους στο ίδιο καλάθι και να πούμε ότι όλα τα προϊόντα του φινικελίου πρέπει να απαγορευτούν. Ό,τι δεν είναι βιώσιμο, ναι, να κηρυχθεί εκτός νόμου. Ε. Διακόπτη πρόεδρος, μάλιστα. Καλά, νομίζω ότι απάντησα πολλές ερωτήσεις. Αυτά. Σας ευχαριστώ. Ό,τι δεν σας ε, απάντησα ε, μπορεί να σας καλύψουν οι συνεργάτες μου. Ελάτε σε επαφή μαζί τους. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε, λέει πρώτα. Σας ευχαριστούμε για όλες αυτές τις ερωτήσεις που απαντήσατε. γραπτές απαντήσεις όποιος χρειάζεται θα λάβει. Στις 13 Μαρτίου η επόμενη συνεδρία. Ευχαριστούμε.